Mesdames, Κυρίες και κύριοι, σας προτείνω να επαναληφθεί η συνεδρίαση. Σήμερα το πρωί θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων ε, με εκπροσώπους της Ανδόρας, Λίχτενστάιν και του ε, Μονακό με αλφαβητική σειρά. ορίζω τους εκπροσώπους και τους χαιρετώ. Θα ε, ακολουθήσουμε μια ελαφρώς διαφορετική διαδικασία από τη χθεσινή, διότι χτες Είχαμε δύο δίκαιοδοσίε και μάλιστα δίδυμε: Γκένζε και Τζέρζι. Οπότε μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο να τους αντιμετωπίσουμε ως ένα συνομιλητή. Τώρα έχουμε τρεις διαφορετικούς συνομιλητές που έχουν ε, κοινά στοιχεία. Είναι πριγκιπάτα κυρίαρχα, ε, δεν υπόκεινται στο βρετανικό στέμα Ορισμένα μάλιστα έχουν και νομικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ως διαδικασία λοιπόν θα ζητήσουμε από κάθε εκπρόσωπο των τριών ε, πριν κυπάτων να κάνει μια εισαγωγική παρατήρηση 7 λεπτή, 8 λεπτή το πολύ. Θα σας ήμουν ευγνώμων να αντιρρήσετε αυτό το χρόνο για να δούμε πώς έχει η φορολογική κατάσταση, το καθεστώς και οι αλλαγές που γίνονται αυτόν τον καιρό στις δικαιοδοσίες αυτές και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο σε όλους τους εγγεγραμμένους ομιλητές ομαδοποιώντας ε, τις ερωτήσεις, τέσσερις βουλευτές κάθε φορά για να γίνει μια ζωηρή και επικοδομητική όσο γίνεται η συζήτηση. Με αλφαβητική σειρά θα δώσω πρώτα το λόγο στην εκπρόσωπο της, οχ, δημοκρατίας πρέπει να πω, ε, του πριγκιπάτου της Ανδόρας cest a euh, Είναι η κυρία Κλάουδια Τονέρα Ντουράνη, που είναι υφυπουργό για τι διεθνεί οικονομικέ σχέσει. Καλημέρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. For Είναι τιμή για την Ανδόρα αυτή η πρόσκληση να παρουσιαστεί στην Επιτροπή σας Πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον ε, να έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψει και να συζητήσουμε τι ε, ιδιαιτερότητε Ανδόρα όσον αφορά τι πρόσφατε εξελίξει, όσον αφορά τη φορολόγηση επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω και όσα για θέματα φοροδιαφυγή, ανταλλαγή πληροφοριών και διάβρωση φορολογητέ ε, βάση. Σχετικά με αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι η Ανδόρα ξεκίνησε μια διαδικασία μεταρρύθμιση εδώ και κάποια χρόνια, από το 2009 και θέλει να πετύχει διαφάνεια σύμφωνα με διεθνεί προδιαγραφέ ανταλλαγέ πληροφοριών και να εξηγιανθεί το ρυθμιστικό μα πλαίσιο, το οικονομικό και το φορολογικό. Θέλουμε να υιοθετήσουμε τι διεθνεί προδιαγραφέ του ΩΣΑ. Υπογράψαμε διάφορε συμφωνίε για ανταλλαγή πληροφοριών τα φορολογικά και ξεκίνησε η προσπάθεια με τη δικήρυξη των Παρισίων τη 10η Μαρτίου του 2009. Εκεί εκφράσαμε τι προθέσει μα να δρομολογήσουμε διαδικασία νομοθετικών μεταρρυθμίσεων του τραπεζικού απορρίτου για να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικών κατόπιν αιτήματο. δυνάμει το άρθρο 26 τη συμβάσεω του ΟΣΑ. Μέχρι τώρα έχουμε υπογράψει 24 συμφωνίε για ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικά ε, με τις εξής δικαιοδοσίες Αυστρία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Άγιος Μαρίνος, Γαλλία, Βέλγιο, Αργεντινή, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ισλανδία, Φιλανδία, νήσι Φερόε, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γρυλανδία, Γερμανία, Αυστραλία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Ελβετία, Κορέα και Ιταλία και επιπλέον έχουμε συνομιλίες με την Νότια Αφρική και τη Σλοβακία. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας 2011-2015 η κυβέρνηση ήδη δρομολόγησε ένα άνοιγμα της οικονομίας μας. Στόχος να ανοίξουμε νέες αγορές και να έχουμε ποικιλομορφία όσον αφορά την οικονομία μας. Πριν από αυτό η αγορά της Ανδόρας δεν ήταν ανοιχτή σε ξένες επενδύσεις και υπήρχε μια οικονομική απομόνωση επιζήμια για τη χώρα, βλέποντας και ποια ήταν και η γενική κατάσταση, η ύφεση. Γι' αυτό το 2012 αποφασίστηκε να αρθούν οι περιορισμοί για τις ξένες επενδύσεις και να επιτρέψουμε σε ξένη συμμετοχή μέχρι 100% του κεφαλαίου επιχειρήσεων και να έχουν δικαιώματα όλοι κάτι και από την πρώτη ημέρα διαμονής. Θέλαμε να διευκολύνουμε ε, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και αγορών, εστιαζόμενοι κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών. Το οικονομικό άνοιγμα δεν αρκούσε. Έπρεπε να προωθήσουμε ένα φορολογικό μοντέλο που είναι συγκρίσιμο και ανταγωνιστικό. Μια φορολογική πολιτική που θα μπορεί να συνδέσει την Ανδόρα με τους γείτονές της. Και γι' αυτό την περασμένη ε, θητεία θέλαμε να αλλάξουμε το φορολογικό μοντέλο της Ανδόρας που θεωρείται ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση. Ένα πλαίσιο είχαμε για τους πολίτες, ενεκρίθη αυτό τον Απρίλιο του 2014 και τέθησε ισχύ τον 1η Ιανουαρίου του 2015 και όσον αφορά τους άλλους νέους νόμους περιφορολογήσεων, οι μη κάτοικοι ε, καλύπτονται από νομοθεσία του 2011. Φόρος εταιριών και οικονομικών δραστηριοτήτων ετέθησαν σε ισχύ την 1η του 2012 και ο νόμος για το ΦΠΑ ετέθησε σε ισχύ την 1η Πρώτου 2013. Το φορολογικό σύστημα της Ανδόρας έχει 10% άμεση φορολόγηση, φορολογικού συντελεστή και 4,5% έμεση φορολόγηση. Το μοντέλο αυτό είναι ενεκρίθη ήδη από τι πρώτε χώρε με τι οποίε κάναμε διαπραγματεύσει για συμφωνίε διπλή φορολόγηση. Τα DTAs που θα λέμε από εδώ και πέρα. Για να αποφευθεί η διπλή φορολόγηση. Μέχρι τώρα η Ανδόρα έχει υπογράψει συμφωνίε τέτοιε με τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Λίχτενστάιν και τα Εμμυράτα και έχει ξεκίνησει διαπραγματεύσει για συμφωνία με τη Μάλτα για αποφυγή διπλή φορολόγηση. Εξακολουθεί να επεκτείνει το δίκτυο τη ε, όσον αφορά τι συμφωνίε αυτέ. Θα, επιτρα... θα, θα μπορούμε να εξάγουμε υπηρεσίε από εταιρείε τη Ανδόρα προ το εξωτερικό χωρί να έχουν φορολογικό επιβάση. Η υπογραφή των συμφωνιών σημαίνει ότι ακολουθούμε σωστό δρόμο όσον αφορά το άνοιγμα τη αγορά χωρί εξαιρέσει και έτσι θα ανοίξουμε προ τα έξω την αγορά μα. Η Ανδόρα συνεργάζεται με άλλε χώρε για να πετύχει νέε τέτοιε συμφωνίε για αποφυγή διπλή φορολόγηση. Το οικονομικό άνοιγμα και εφαρμογή ενό φορολογικού μοντέλου που είναι συγκρίσιμο και ανταγωνιστικό και διαπραγματεύσει των συμφωνιών με μη διπλή φορολόγηση δημιουργούν ελκυστικό περιβάλλον και μια σύγχρονη οικονομία για τη χώρα. Η Ανδόρα έχει πολύ σημαντικό εμπορικό και τουριστικό τομέα. Περίπου 8 εκατομμύρια επισκέπτε το χρόνο έχουμε. Εκατό φορές περισσότεροι οι τουρίστες έρχονται από τους μόνιμους κατοίκους. Το κλίμα αυτό επιτρέπει να αντιθούν και άλλοι τομείς, όπως η υγεία, η παιδεία και η νέα τεχνολογία που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού και του εμπορίου. Ποια είναι η ιδέα. Οι νέοι τομείς εποφελούνται από το εμπορικό και τουριστικό δίκτυο τη Ανδόρα για να αναπτύξουμε προϊόντα και υπηρεσίε. Και αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίε βοηθούμε να πετύχουμε ισορροπία μεταξύ των παθησικών τομέων τη χώρα και τη ανάπτυξη νέων οικονομικών μοντέλων οριζοντας 2013 2013-2020 υπογράψαν συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιούμε το ευρώ σαν επίσημο νόμισμα και μπορούμε να έχουμε και ε, νομίσματα που κόβουμε ευρώ. Και πρέπει να εφαρμόσουμε επίσης και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την πρόληψη νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων, να μην έχουμε παραποίηση, παραχάραξη το ευρώ. Έχουμε κανόνες για τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα σε ευρώ και κάποιου χρηματοπιστωτικού κανονισμούς ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζουμε άμεσα σύμφωνα με προθεσμία που προβλέπεται για την ενσωμάτωση των νομοθεσιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη δική μα αναμετάξη. Από τον Απρίλιο 2012 υπογράψαμε τη Ευρωπαϊκή Συμφωνία και την εφαρμόσαμε. Το νομικό πλαίσιο τροποποιήθηκε για να προσαρμοστεί στι νομικέ πράξει και ρυθμιστικέ διατάξει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, όπω αναφέρονται ε, στο παράτημα τη Συμφωνία του Νομισματικά. Το περασμένο Οκτώβριο στην Ανδώρα έγινε η τέταρτη συνάντηση τη Μικτή Επιτροπή τη Νομισματική Συμφωνία. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι μέχρι τώρα η έγκριση του πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στην Νομισματική Συμφωνία γίνεται εντό τη προθεσμία που προβλέπετε Και ο τρόπο δείχνει ότι είναι αξιόπιστη η ανδώρα και ότι είναι σοβαρή και ότι σέβεται τι υποχρεώσει που έχει αναλάβει. Παρ' όλα αυτά όμω θέλουμε να σα πούμε ότι η Ανδώρα ανησυχεί πάρα πολύ διότι θεωρείται ότι είναι μια δικαιοδοσία ότι δεν συνεργάζεται πλήρω ή φορολογικό παράδεισο θεωρείται. τελευταία χρόνια θεωρούμε ότι δείξαμε στον κόσμο ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ανδόρα όλα τα θέματα που αφορούν την οικονομική διαφάνεια και την ορθή διακυβέρνηση να τα εφαρμόζουμε. Πραγματι έχουμε δεσμευτεί έναντι Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΣΑ να συμμορφωθούμε με τι παγκόσμιε προδιαγραφέ του ΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα φορολογικά. Το 2011 ήδη συμφωνήσαμε και κάναμε σημαντικά βήματα τόσο ώστε να πετύχουμε τον λόγο στόχο. Συμμετεί, συμμετέχει η Ανδόρα στο Παγκόσμιο ε, Φόρουμ στην ομάδα υψηλού επίπεδου. Θα παριθμίσω κάποιες βασικές δράσεις που έχει δρομολογήσει η Ανδόρα. 5 Νοεμβρίου του 2013 η κυβέρνηση της Ανδόρα υπέγραψε τη σύμβαση για αμοιβαία διοικητική αρρωγή για τα φορολογικά με τον ΩΣΑ. Περιμένουμε να εγκυρωθεί κατά το πρώτο εξάμεινο του 2016 Στι 16 Ιουνίου του 2014 Ιουνίου υιοθέτησε τη δήλωση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από τον ΟΣΑ και έγινε η 48η δικαιοδοσία που συμμορφώθηκε με τις προδιαγραφέ σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητα. Στις 3 Δεκεμβρίου του 2015 η Ανδόρα επέγραψε την πολυμερή συμφωνία για τον αρμοδίων αρχών και έγινε η 75η δικαιοδοσία που το επέγραψε αυτό. Υπέχει υποχρέωση να εφαρμόσει ενίο πρόγραμμα ανταλλαγή πληροφοριών, κάτι που προβλέπεται από τον ΟΣΑ. Στις 12 Φεβρουαρίου του 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ανδόρα υπέγραψαν ένα κείμενο για μια νέα συμφωνία για διαφάνεια τα ε, που είχε μονογραφηθεί στις 4 Νοεμβρίου του 2015. Σύμφωνα με την Νέα Συμφωνία, η Ανδώρα και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αυτομάτως ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τους οικονομικούς λογαριασμούς των κατοίκων τους από το 2011 και πέρα. Αυτή η συμφωνία ανανεώνει και τροποποιεί τη συμφωνία που υπεγράφει το 2004 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ανδώρας όσον αφορά τη θέσπιση μέτρων που αντιστοιχούν με αυτού που αναφέρονται στην οδηγία 2003 κάθετο 48 κάθετο ΕΟΚ όσον αφορά τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων ε, ε, υπό τη μορφή πληρωμών τόκων. Συμμετείχε στη δημιουργία της ομάδας του πολυμερούς ε, εργαλείου του ΟΣΑ και συμμετέχουν στη κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε και να συμμορφωνόμαστε με του διεθνεί κανόνε. Γι' αυτό ξεκινήσαμε διαπραγματεύσει για τη Συμφωνία Συνδέσεω με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά αυτή την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να σημειώσουμε ότι στι 18 Μαρτίου του 2015 ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ανδόρα συμμετείχε στι Βρυξέλλε σε επίσημο γεύμα των διαπραγματευτών ε, και συζήτησαν μία, δύο περισσότερες ε, για τη συμφωνίες συνδέσεις μεταξύ ε, Ανδόρας, ε, Αγίου Μαρίνου και Μονακό. Αν μπορείτε να συντομεύετε, λέει ο Πρόεδρο. Κλείνοντα, θα θέλω να πω ότι η πολιτική προτεραιότητα τη κυβερνήσεω του Πριγκιπάτου τη Ανδόρα είναι η χώρα να γίνει όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Από αυτή την έποψη, εξυγίανση του φορολογικού και οικονομικού ε, πλαισίου είναι βασικό κλειδί για την κυβερνητική πολιτική. Αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο που συνδέεται με την πρόθεση τη κυβερνήσεω να αντισταθμίσει, να εξισορροπήσει τα δημοσιονομικά, θέλει να κάνει μια χώρα που είναι ελκυστική, ανοιχτή, ανταγωνιστική, παγκοσμιοποιημένη και επίση συμφωνεί με διεθνεί η Ανδόρα δεν παραμείνει ε, κολλημένη στο παρελθόν και γι' αυτό η κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει να ανοίξει τον κόσμο ώστε να αυξηθεί η οικονομία μας, να αναπτυχθεί. Και θα πρέπει όλα να ελέγχονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές για περί διαφανείας και να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το νομικό πλαίσιο και να έχουμε ισότιμε συνθήκε με στην μικρή χώρα που πρέπει να διατηρήσει ανταγωνιστικό μοντέλο, επιτρέποντα όμω κάποιε ιδιαιτερότητε να είναι ελκυστικέ. Με όλε αυτέ τι θαραλέε και αναγκαίε μεταρρυθμίσει, η Ανδώρα ε, είναι μια χώρα που είναι έτοιμη να αναπτυχθεί μια ανάπτυξη που δεν θέλουμε, μια χώρα που δεν θέλουμε να είναι απομονωμένη και να είναι μια εξαίρεση, να είναι αποτέλεσμα σχέσεων μεταξύ Ανδόρα και των γειτονικών χώρων. Να μην αναπτύσσεται μόνο λόγω ιδιαιτεροτήτων, λόγω συνεργασία. Ευχαριστώ. Θυμίζω το εξή. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών που υπεγράφει στι 12 Φεβρουαρίου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία αυτή προσεχώς θα υποβληθεί προς έγκριση στο Συμβούλιο Υπουργών αφού θα έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλλον ήδη εγκρίθηκε στην περασμένη μας ε, σύνοδο. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Κάτια Γκέι, έτσι προφέρεται. Γκάι, μάλιστα. Ζητώ συγγνώμη. Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνών Οικονομικών Υποθέσεων στο Λίχτενστάιν. Οκτώ λεπτά παρακαλώ αν μπορείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δίνετε την ευκαιρία στο Λίχτενστάιν να παρουσιάσει τη θέση του σε σχέση με τις θέσεις της εξελίξης σε επίπεδο ΕΕ και ΩΣΑ για την διαφάνεια ανταλλαγή πληροφοριών και διάβρωση τη βάση και μετατόπιση κερδών. Ε, είναι βασική εταίρη μα ε, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στα πλαίσια μόνο τη κοινή ενιαία αγορά, γιατί εδώ και πάνω από 20 χρόνια συμμετέχουμε σε αυτά και πέραν αυτού ε, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά και γι' αυτό καλωσορίζουμε οποιαδήποτε πρόσκληση για εμβαθμένο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με υπόλοιπα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο με χαρά θα ανταλλάξουμε τις ε, απόψεις για, κυρίως για τόσο σημαντικά ζητήματα όπως η φορολόγηση. Προτού περάσω στο αντικείμενο της ανταλλαγής απόψεων θα ήθελα να σας δώσω και κάποιες γενικές πληροφορίες για το Liechtenstein. Ναι, θα ήθελα έτσι να διευκρινίσω κάποια πράγματα και να συμπληρώσω την εικόνα που έχετε για το Liechtenstein δεν θεωρείται τόσο συχνά ως φορολογικός παράδεισος ή ούτε είναι η ειδική φορολογική δικαιοδοσία ούτε η οικονομία βασίζεται μόνο σε παροχή υπηρεσιών ή έχει σε ένα μόνο οικονομικό κέντρο. Το Λίχτενστάιν ιδρύθηκε πριν από πάνω από τρει αιώνε ε, και ε, έχει διαφυλάξει την εθνική του κυριαρχία. Βρίσκεται στην καρδιά τη Ευρώπη ε, και είμαστε από τι πλέον ανεπτυγμένε κοινοτόμε περιοχέ ανάμεσα στην Ελβετία, την Αυστρία και την Νότια Γερμανία είναι εξαιρετικά καινοτόμο ο παραγωγικός και μεταποιητικό μα τομέα που συμβάλλει στο 40% τη οικονομία μα Σε κατακεφαλή για το Λίχτενσαν μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι είμαστε από τι πλέον βιομηχανοποιημένε χώρε, όχι μόνο τη Ευρώπη, αλλά και του κόσμου ε, με ένα ποσοστό επιχειρηματικότητα κατακεφαλή που μα κάνει περήφανου. Ε, Γεφύρες, κτίρια, να τον κόσμο κατασκευάζονται με υλικά που προέρχονται από το Λίχτενσταν. Η θέρμανσή σα μπορεί να προέρχεται από το αυτοκίνητό σα κατά πάσα πιθανότητα έχει συστήματα οδήγησης και χρησιμοποιεί συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στο ε, Λίχτενστάιν. Ε, το μικρόφωνο σας ε, παραδείγματο χάρη χρησιμοποιεί ένα εξάρτημα από εταιρεία μας που έχει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμια κλίμακα, όπως και άλλες εταιρείες μας ε, και κυρίως σε μικρά τμήματα της αγοράς, θα λεγόμενα νης. Οι οικονομικές υπηρεσίες αντιστοιχούν στο 24% του ΑΕΠ μας ε, και το υπόλοιπο είναι άλλες λοιπές υπηρεσίες ε, και γεωργικός τομέα. Συνολικά για την οικονομία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στο χρηματοπιστωτικό ταμείο. Έχουμε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, επενδυτικές εταιρείες, ε, έχουμε πολύ καλή κεφαλαιοποίηση στι τράπεζες ε, του Λίχνεστάιν ε, και κατά τη διάρκεια τη παγκόσμια χρηματοπιστωτικής και στο 2008 δεν χρειαστήκαν στήριξη. Συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο από το 1995 και μετά και Επιλέξαμε το, συνειδητά τον δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ως απόρρια μιας ε, ε, άμεσα δημοκρατικής ε, διαδικασίας διαβούλευσης με τους πολίτες. Μέσα από αυτή την συμφωνία του ΕΟΧ μαζί με την Ισλανδία το Λίχτενστάιν συμμετέχει στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώντας έτσι τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Τι σημαίνει αυτό. Το Λίχτενστάιν πρέπει το, το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το μεταφέρει ακέραιο ε, στην εσωτερική ένωμη τάξη. Όλοι οι κανονισμοί, όλες οι οδηγίες για τις χρηματοπιστικές υπηρεσίες ως εκ τούτου, καθώς και για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών και διατάξεις για την καταπολέμηση της, ε, του ξεπλήματος χρήματος νομιμοποίησης, δηλαδή παρανόμων εσόδων, υποχρεώσεις αποκάλυψης, ε, όλο το, το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται ήδη στο Λίχτενστάιν. Πριν από 10 χρόνια περίπου, ε, λάβαμε μια πολύ σημαντική απόφαση με σημαντικότατες επιπτώσεις ε, το 2008 και 2013 με δηλώσει η κυβέρνηση επιβεβαιώθηκε αυτό και ο στόχο ήταν να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές μας σε διεθνές επίπεδο για συνεργασία σε φορολογικά ζητήματα. Αυτή η απόφαση για την πολιτική μας βασίζεται στην γνώση που έχουμε ότι πλέαρα από αυτές τις κοινέ αξίες και το κοινό και εκτιμένο βασιζόμαστε και σε χρηματοψηφιακές αγορές για την βιομηχανία μας και τις υπηρεσίες μας. Έκτοτε λοιπόν το Λίχτενστάιν ενστενίστηκε πλήρω και όχι μόνο, αλλά συνέβαλε στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων προ τη διαφάνεια για τα φορολογικά ζητήματα και τη συνεργασία σε αυτά. Ε, πρόκειται λοιπόν ε, για μια συνολική προσέγγιση που ε, με προορατικό τρόπο και με ιδιαίτερη συνέπεια εφαρμόζεται έκτοτε στην νομοθεσία μας και στον ακρονιστικό μας πλαίσιο. Το 2010 το Λίχτενστάιν αναθεώρησε άρδινε το φορολογικό του σύστημα. Ο στόχος ήταν να επιτύχουμε ουδετερότητα ως προς τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα με αυτή τη μεταρρύθμιση ο εταιρικός φόρος του Λίχτενστάιν προσαρμόστηκε στις διεθνείς και ευρωπαϊκές ευρωπαϊκές εξελίξεις καθώς και στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Συμβατότητα με την ε, τέσσερις βασικές ελευθερίες ε, και τις ε, διατάξεις της κρατικής κρατικές ήταν κινητήριος δύναμη της μεταρρύθμισης, αποφυγή μέτρων ring fencing και ειδικών λογικών καθεστώτων. Τώρα υπάρχει ε, ένας, ε, ένας ε, καθολικός συντελεστής 12,5% για τις εταιρείε. Εφαρμόζουμε την αρχή arm's length και τις κατευθύνες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τα εισοδήματα που έχουν ανά τον κόσμο φορολογούνται οι εταιρείε και χρησιμοποιούμε προοδευτικούς φορολογικούς συντελεστές. Ο οριακός συντελεστής φτάνει μέχρι και 24%. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι το Λίχτενστάιν έχει ήδη υποβάλει σημαντικά της φορολογικής του νομοθεσίας μέσα στις ε, εποπτικές αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το πώς να ε, ε, ισχύουν. Αυτό είναι το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι, για τον ΕΟΧ και έχει αρμοδιότητα την επόπτευση και την εφαρμογή των υποχρεώσεων της Συμφωνίας ΕΟΧ. Αυτό σημαίνει όλων, όλου του εφαρμοστέου δικαίου στις τρεις χώρες ΕΟΧΕΖΕΣ. Ε, έτσι η ΕΣΑ, η Εποπτική Αρχή, ε, ενέκρινε μεταξύ άλλων το box για τα πνευματικά δικαιώματα και λοιπά κομμάτια του φορολογικού γεκτημένου του Λιχτενστάιν. Επίσης αναθεωρήθηκε η πρακτική μας για τις φορολογικές συμφωνίες tax ruling και ε, μετά την αξιολόγηση κρίθηκε ότι συνάδει με την κείμενη νομοθεσία και δεν περιέχει επουδενή κρατικές ε, ε, επιδοτήσεις. Τώρα, Εντάχει να δούμε τη θέση του Λιχτεστάνη για τα φορολογικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματο ε, και σε συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη. Το Λίχτενστάιν ε, διαθέτει ένα καθολικό δίκτυο διμερών αλλά και πολυμερών συμβάσεων ε, με τις τελευταίες εξελίξεις ως προς τις διατάξεις για τις κρατικές επιδοτήσεις. Έχουμε κριθεί ως συμμορφούμενοι με το παγκόσμιο κεκτημένο από χώρες όπως η Ολλανδία και η Ιταλία παραδείγματο χάρη σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε επιτύχει από παγκόσμιους φορείς θετική αξιολόγηση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αναφερθήκατε και εσείς σε αυτό. Ε, ε, ε, ήδη πάρα πολύ νωρίς υποστηρίξαμε τα νέα πρότυπα, τα εγκρίναμε και τα εφαρμόσαμε και παραδείγματο χάρη η συμφωνία για την εφορολόγηση των αποταμιεύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση βασιστήκαμε στο χρονοδιάγραμμα που άρχισε να ισχύει ήδη την πρώτη πρώτου. Επίσης για την εφαρμογή της νομοθεσίας μπορούμε να πούμε ότι είναι εφαρμοστές ήδη οι σχετικές διατάξεις. Τώρα για τον τον υγιή φορολογικό Ταγωνισμό και τις αθέμενε φορολογικέ πρακτικές, το Liechtenstein ε, ακολουθεί τα πρότυπα BEPS του όσα Έχουμε αρχίσει να αναπτύσσουμε τα απαιτούμενα μέτρα για την φορολογική πολιτική ε, που σχετίζεται με το BEPS για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε σωστά τα πρότυπα. Επίσης υπογράψαμε ε, πολυμερή συμφωνία για τις αρμόδιες αρχές για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα. Council Reporting και έχουμε αρχίσει διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του κώδικα διοντολογίας για τη φορολόγηση των εταιριών το 2010 κατά πάσα πιθανότητα. Ε, στον επόμενο γύρο θα μπορούσα να επεκταθώ ε, για αυτά τα ζητήματα που σας απασχολούν. Διακόψαμε ε, για ένα χρονικό διάστημα αυτό το διάλογο και ε, πρόσφατα το 2014 συνεχίστηκε επί τη βάση ενός, μιας προσέγγισης roadmap, δικού χάρτη. Πιστεύουμε πως ε, αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να βασίζεται σε ισότιμους όρους και έχουμε κάθε πρόθεση να συζητήσουμε τα θέματα που έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση Ταυτόχρονα όμω θα θέλαμε να συζητήσουμε και θέματα που μας απασχολούν και εμά. Εν κατακλείδη, Πρόεδρε, με τα χαράς να συζητήσουμε, να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις και να τονίσω ότι θα εξακολουθήσουμε να είμαστε επικοδομητικοί ε, εταιροί για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τα κράτη-μέλη. Πρώτα, σας ευχαριστούμε κύριε μου. Χαιρόμαστε όλους ιδιαίτερους που μαθαίνουμε ότι είναι βιομηχανική δύναμη το Λιχτενστάιν ορισμένε φορέ υποτιμούμε τη σημασία του τομέα αυτού. Θα επανέλθουμε στο θέμα των λαϊκών συμφωνίων. Από τα πριγκιπάτα, το Λιχτεστάιν ήταν πρώτο που στι 28 Οκτωβρίου 2014 σύναψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανταλλαγή φορολογικών δεδομένων. Η συμφωνία ετέθη ισχύ μετά την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου και την ε, απόφαση του Κοινοβουλίου στις 8 Δεκεμβρίου του 2014. Πριγκιπά το Μονακό, ο ο κύριο Ζαν Καστελίνη, Υπουργό Σύμβουλο της Κυβέρνησης για Φορολογικά Ζητήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Πριν από ένα μήνα και λιγότερο είχα τη χαρά να ε, μονογράψω παρουσία του ε, Επιτρόπου Μοσκοβισή το πρωτόκολλο τροποποίησης συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό που προβλέπει ε, μέσα για την οδηγία 2003 48 του Συμβουλίου. Αυτή η μονογραφή είναι πολύ σημαντική στα πλαίσια της πολιτικής του Μονακό για την καταπολέμηση της διεθνούς και φοροδιαφυγής. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε ότι εγγράφεται ως συνέχεια της προσπάθειας και της δέσμευσης ε, που ε, έχει αναλάβει ε, ο γαλινότατος πρίγκιπς Αλβέρτος δεύτερος τα τελευταία χρόνια. Έχουμε διμερείς και πολυμερείς συμβάσεις και συμφωνίες για ανταλλαγή πληροφοριών, διεθνές προδιαγραφές. Σεβόμαστε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκοσμίου Φόρουμ του ΟΣΑ και ε, χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χαρακτηρίζουν ότι συμμορφωνόμαστε σε μεγάλο βαθμό. Εδώ και δύο και πλέον τι έχουμε διαπραγματεύσεις ε, δική μας αντιπροσωπεία με την Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα με ε, την ε, Ελβετική Συνομοσπονδία, το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, το Πριγκιπάτο του Λίχτενστάιν και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου. Αυτές οι διμερείς διαπραγματεύσεις καταλήγουν σε ένα κείμενο που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Μονακό, βεβαίως η συμμεταχείριση πάντα με τις άλλες τρίτες χώρες και τις αντίστοιχες συμφωνίες. Αυτές οι ιδιαιτερότητες είναι εκ των όνων κάνευ για το Μονακό. Για να διαφυλάξουμε την καλή μας οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση και το βιωτικό μας επίπεδο και από αυτό εξαρτάται κατά κύριο λόγο και πρώτο λόγο η κυριαρχία μας και κατά δεύτερο λόγο η ένταξή μας στον κόσμο. Αυτή η ευρωστία οικονομική και χρηματοπιστωτική επέτρεψε στο πριγκιπάτο μας να μην δανείζεται. Ε, το 2015 έχουμε ένα οικονομικό έτος που είναι η τέταρτη συνεχής ε, ε, χρονιά σε πλεόνασμα και ο αρχικός προϋπολογισμός του 2016 έχει ψηφιστεί επίσης πλεονασματικός. Αυτό το αποτέλεσμα βασίζεται στη συμμετοχή όλων των κλάδων της οικονομίας, του Μονακό και ιδιαίτερα ε, του βιομηχανικού μας ιστού. Προσπαθούμε να ε, προσαρμοστούμε στον εξωτερικό κόσμο και να παραμένουμε ελκυστικοί για τους οικονομικούς παραγόντες παγκοσμίω. Κάθε τομέα έχει τη σημασία του, αντίστοιχη και συγκρίσιμη, γιατί μία από τις ισχύες, ε, τις δυνάμεις μας είναι αυτή η ποικιλομορφία και διαφοροποίηση. Δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις μας και σε μεγάλο βαθμό από εκεί ε, προέρχονται τα φορολογικά μας έσοδα και θα επανέλθω σε αυτό. Και παρά τη διεθνή κρίση καταφέραμε να προσελκύσουμε όλο και περισσότερους μόνιμους κατοίκους και επενδυτές τα τελευταία χρόνια. Έχει μια διεθνή ακτινοβολία το Μονακό την οποία συχνά και θετικά αξιολογούν και χαιρετίζουν και οι δύο γείτονε μας η Γαλλία και η Ιταλία ε, όπου η οικονομία μας παρέχει ε, χιλιάδες ε, θέσεις εργασίας. 45.000 εργαζόμενους έχουμε από την Ιταλία και τη Γαλλία σε 5.000 επιχειρήσεις στο Μονακό. Και δύο είναι βιομηχανικές επιχειρήσεις και ο επίτροπο Μοσκοβισή είχε την ευκαιρία να τι επισκεφθεί όταν μετέβη στο πριγκιπάτο του Μονακό. Άρα... Βέβαια σήμερα μας απασχολεί ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων ε, και γι' αυτό θα ήθελα να σα δώσω κάποια τεχνικά στοιχεία για το πώς φορολογούνται οι ε, επιχειρήσεις στο Μονακό. Υπάρχει φόρο στα κέρδη, φόρο στο στιθέμενη αξία και ε, φόρος ε, τέλος καταχώρηση. Και έχουμε συνεργασία στενή με τη Γαλλία, με συμβάσεις που διέπουν τις ε, δύο χώρες 18 Μαΐου 1963 ε, για θέματα δασμολογικά και φορολογικά και ορίζει ότι η Γαλλική και ε, επικράτεια του Μονακό έχουν τελωνιακή ένωση. Άρα ο τελωνιακός κώδικα, οι δασμοί εισαγωγικών και εξαγωγών, καθώς επίσης και οι άλλοι δασμοί που αφορούν τη Γαλλική Δημοκρατία, βρίσκουν εφαρμογή και στο πριγκιπάτο του Μονακό. Ε, για τη φορολογία τώρα η συμφωνία επιβάλλει φόρο επί των κερδών και ο φόρος προστιθέμενης αξίας ε, είναι στην ίδια βάση και με τον ίδιο φορολογικό συντελεστή όπως και στη Γαλλία. Σε ό,τι αφορά το φόρο επί των κερδών, το πρώτο άρθρο αυτής της φορολογικής σύμβασης ορίζει ότι με επιφύλαξη των ε, περαιτέρω προσαρμογών που θα χρειαστούν λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης του πριγκιπάτου, ο φόρος αυτός ε, συλλέγεται και καθορίζεται με τους ίδιους όρους όπως και ο γαλλικός φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων. Έτσι, ε, υπόκεινται σε αυτό το φόρο οι εταιρείε ανεξαρτήτως μορφής, φυσικό νομικό πρόσωπο που ε, έχουν βιομηχανική εμπορική δραστηριότητα στην επικράτεια και όταν ο κύκλος εργασιών από 25% τουλάχιστον προέρχονται από άμεση ή έμεση δραστηριότητα. 33,33% ε, είναι ο φόρος επί των κερδών ε, σε ένα οικονομικό έτος και μετά φόρου από όλες τις δραστηριότητες ε, που ασκούν οι επιχειρήσεις. Ό,τι αφορά το ΦΠΑ, έχουμε το άρθρο 15 της Φορολογικής Σύμβασης που σας προανέφερα και το άρθρο 7 της Οδηγίας 2006-112 ε, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φόρο προσθέμενης αξίας. Για το άρθρο 15 της Σύμβασης 18 Μαΐου του 1963 ορίζει ότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας στο Μονακό επιβάλλεται με τους ίδιους όρους και με τον ίδιο φορολογικό συντελεστή όπως και στη Γαλλία. Έτσι λοιπόν με κυρίαρχα διατάγματα μεταφέρει στην εσωτερική ένωμη τάξη το Μονακό ε, τις διατάξεις περί ΦΠΑ που ε, ε, συμπεριλαμβάνονται στο φορολογικό νόμο της Γαλλίας και στα αντίστοιχα διατάγματα. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 7 της οδηγίας που σας προανέφερα, προβλέπει αυτή ότι ε, λόγω των ε, σχέσεων και των συμβάσεων που έχουμε προσυπογράψει με τη Γαλλία δεν θεωρείται τρίτη χώρα για την εφαρμογή της οδηγίας αυτή στο Μονακό αλλά εξισώνεται με τη Γαλλία και ε, το καθεστώς ε, το φορολογικό για το ΦΠΑ που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει και στο Μοναχό και οι πολίτες που διακινούν αγαθά ή υπηρεσίες έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με εκείνους που φορολογούνται στη Γαλλία. Σε ό,τι αφορά το τέλος καταχώρησης της εταιρεία, η υπηρεσιες εχουν τις ιδιες υποχρεωσεις με εκεινους που φορολογουνται στη γαλλια σε οτι αφορα το τελος καταχώρηση τη εταιρεια η νομοθεσια μας ε, ε, βασίζεται ε, στη λειτουργία της επιχείρησης 1% για την αύξηση κεφαλαίου για τα συμβόλαια για την εκχώρηση μεριδίων ή μετοχών και 7,5% για το τον αέρα μια επιχείρηση. Τα φορολογικά έσοδα από τις επιχειρήσεις ε, είναι ο βασικός όγκος ε, των εσόδων του προπολογισμού του κράτους μας. Οι φόροι λοιπόν επί των κερδών και ο ΦΠΑ το 2015 είναι το 78 περίπου της 100 των ετησίων φορολογικών εσόδων και 60% του ε, προϋπολογισμού του κράτους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Βάλατε στο σύνολο και το ΦΠΑ που καταβάλουν οι επιχειρήσει. Καλώς σας ευχαριστώ. <laughs> Πρώτες ρηπέ ερωτήσω. <laughs> Ε, να διευκρινίσω κάτι με το Μονακό. Όπως αναφέρατε κύριε Υπουργέ, ολοκληρώνται οι διαπραγματεύσεις. Η υπογραφή προβλέπεται Απρίλιο. και έγκρισε το Κοινοβούλιο θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Ο κύριος Γεπ Κόφοντ, ο συνεισηγητής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ανδόρα, το Λίχτενστάν και το Μονακό που ήρθαν στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ για το πνεύμα συνεργασίας που δείξατε για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τα φορολογικά. Το ανέφερε και ο πρόεδρο. Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλό αυτό, είναι πρόοδο. Δείχνει ότι μπορεί να συνεργαστούμε για τη διαφάνεια. Θα επιμείνω από αυτού στη σύντομη παρέμβασή μου. Θα ήθελα λεπτομέρειε. Υποστηρίζετε τι απαιτήσει για τα BEPS του ΟΣΑ όσον αφορά την καταχώρα υποβολή εκθέσεων. Υποστηρίζεται και δημοσιοποίηση των στοιχείων των εκθέσεων κατά χώρα που συζητούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ουσιαστική διοκτησία των εταιριών, των επιχειρήσεων, των καταπιστευμάτων και των ιδρυμάτων. Υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των τριών χωρών. Θα μπορούσατε να εξηγήσετε γιατί δεν έχετε κεντρικό μητρό πραγματικής ιδιοκτησίας και δημοσιοποίηση των στοιχείων. Τέλος. Βλέποντας τους κανονισμούς περί διαφανείας για τα στοιχεία των επιχειρήσεων. Δεν πιστεύω ότι έχετε πλήρη διαφάνεια. Στις πληρωμές αναφέρονται, υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά όλων των πληρωμών και των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα. Μιλάτε για διαφάνεια, μεν, αλλά αν δείτε τα στοιχεία για την πραγματική διοκτησία, την καταχώρα υποβολή εκθέσεων και τους κανονισμούς περί διαφάνεια με τις εταιρείε τις επιχειρήσεις, υπάρχει μεγάλη μυστικότητα, πιστεύω. Μπορείτε εσείς να το σχολιάσετε. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Φρανκ Έγγελ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μικρή μοναρχία από την οποία κατάγομαι από το Λουξεμβούργο. Είναι καλό να συναντώμεθα. Με, να υπάρχουν συναντήσεις μεταξύ του Μεγάλου Δουκάτου και των Πριγκιπάτων. Και έτσι αλλάζει και το ύφος των συνομιλιών. Δύο ερωτήσεις έχω προς εκπροσώπους των τριών χωρών. Πρώτη, Μας ενδιαφέρουν λοιπόν το θέμα των, ε, των φορολογικών για τις αποφάσεις τα φορολογικά, τα tax rulings. Δεν ακούσαμε πολλά για αυτά. Λοιπόν, οι πρακτικές αυτές είναι γνωστές για τις φορολογικές αποφάσεις, για τα tax rulings. Θεωρείτε ότι είναι σημαντικό στοιχείο για την οικονομική σας θέση. Ή είναι πρακτικές που δεν θεωρείται σημαντικές για τις δικές σας διευθετήσεις. Στην αρχή των εργασιών είπε λίγο πολύ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λίγο πολύ α, κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φορολογικός παράδοσος ή κάποιο άλλο. Εμείς στο Λουξεμβούργο αρνούμεθα να χαρακτηριστούμε φορολογικός παράδεισος. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο έχετε όλες, όλοι σχέσεις προνομιούχες θα έλεγα με τους μεγάλους σας γείτονες και υπάρχει πιο άμεση διάδραση με τους διάφορους οικονομικούς φορείς και καταθέτες κάποιων χωρών σε σχέση με άλλες. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Όσον αφορά τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχετε με τις μεγάλες χώρες που συνορεύουν μαζί σας ή με τις χώρες που είναι βασική σας χρηματοπιστωτική και οικονομική εταίρεια. Λοιπόν, αν μπορούσαμε να έχουν παραπάνω λεπτομέρειες γι' αυτό θα μας ευχαριστούσε. Πράγματι, ο Πρόεδρος, είναι μια ερώτηση που θέσαμε χτες στους εκπροσώπους του Γκένσε και του Τζέσε, που έχουν πολύ στενές σχέσεις με κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν του S&D, ο Πίτα Ζήμερα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε πέντε λεπτά για την ερώτηση και την απάντηση, οπότε θα είμαι σύντομος και θα παρακαλούσα να απαντήσουν ένα λεπτό ο καθένα σε τρεις ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Όπως είπε και ο Φωτ, έκθεση αναχώρα. Θα ήθελα συγκεκριμένα να μου πείτε και λεπτομερώς τι σκέφτεστε και αν έχετε την πρόθεση να συμμετέχετε ποιος ε, πληρώνει πόσους φόρους σε ποια χώρα. Ταυτόχρονα θα με ενδιαφέρει να μάθω εάν μπορείτε να φανταστείτε στην ανταλλαγή αυτή πληροφοριών να συμμετέχετε που ε, κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα tax rulings. Δηλαδή τα κράτη-μέλη να έχουν αμοιβαία πληροφόρηση. Και η τρίτη ερώτηση έχει να κάνει ε, με τον, ε, την κοινή ενοποιημένη βάση ε, φορολόγησης επιχειρήσεων που επίκειται. Ε, πώς το βλέπετε αυτό μπορείτε να φανταστείτε να συμμετέχετε σε ένα τέτοιο σύστημα, προτείνετε να νεοθετήσετε τέτοιε ρυθμίσει. Ευχαριστώ, Πέτερ. Από την ECR, αντιπρόεδρο Μπέντ Λούκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχά, έχω ερωτήσει προ το πριγκιπάτο του Λίχτενστάιν και τη Ανδόρα. Ε, για ε, τις ρυθμίσεις ε, της τιμολόγηση των ε, μεταβιβάσεων. Στην Ανδώρα, μάλλον στο Λίχτενστάιν είναι σύμφωνα με ε, ε ανταγωνισμού, το arm's length. Ε, αλλά τι γίνεται με τα κριτήρια και πώς ε, τα μετράτε, για ποιο λόγο δεν δίνονται τα στοιχεία και ε, θα ήσασταν πρόθυμοι να τα διαβιβάζετε. Η εκπρόσωπος του Πριγκιπάτου της Ανδόρας δεν μίλησε καθόλου για αυτό το θέμα. Για τις ε, τιμές των μεταβιβάσεων θα παρακαλούσα να μας πείτε σύμφωνα με ποια αρχή ε, τεκμηριώνονται και ορίζονται. Κατά τα άλλα σύμφωνα και με τις ερωτήσεις του κ. Ζήμων για την ε, ε, κοινή ε, ενοποιημένη φορολογική βάση για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Κυρίως προς το Λεχτενστάιν και την Αντόρα. Και θα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αν πιστεύετε ότι η εισαγωγή μιας τέτοιας φορολογικής βάσης θα ήταν για σας επιζήμια. Σε περίπτωση που θα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα είχε συνέπειες και στα δικά σας φορολογικά έσοδα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Μιγγέλ Βιέγκας από την ΚΟΕ. Καλημέρα. Ανταλλαγή πληροφοριών, αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν είναι τίποτα καινούργιο. Το 2004 εγκρίθηκε μια οδηγία που εφαρμόστηκε το 2005 και Έκτοτε υπήρξε και μια ένα πρώτο κύμα συμφωνιών με κάθε μία από τις χώρες που εκπροσωπούνται στη σημερινή μας συνεδρίαση. Τότε προέκριναν όχι την αυτόματη ανταλλαγή προφοριών εκείνες οι χώρες, αλλά την διατήρηση φόρου ε, επί των επιτοκίων και ε, επί τόκων, και αποφάσισαν ότι θα υπήρξε θα υπήρχε αναδιανομή στους κατέχοντες λογαριασμούς σε αυτές ε, τις δικαιοδοτικές επικράτειες. Βάσει των στοιχείων που έχουμε, τι συνέβη με αυτό το ζήτημα. Πολλές χώρες δήλωσαν ότι δεν έλαβαν ποτέ πληροφορίες, δεδομένα για τους κατόχους λογαριασμών. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι ο απολογισμός αυτής της πρώτης εφαρμογής συμφωνίας το 2005. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε τι έχει αλλάξει έκτοτε και τι μπορεί να μας κάνει να πιστέψουμε ότι αυτές οι αναθεωρημένες πλέον συμφωνίες θα είναι αποτελεσματικότερες ε, εφ' Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στον Ερνέστ Ουρτάσουν, τον συναδελφό μας, γιατί πρέπει να αναχωρήσει σε λίγα λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Η ερώτησή μου είναι προς την Ανδώρα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Απαντώντας στην πρόσκλησή μας, επιμείνετε πάρα πολύ στο γεγονός ότι δεν είστε φορολογικός παράδεισος ή δικαιοδοτική επικράτεια που δεν συνεργάζεται. Επιτρέψτε μας να έχουμε μερικοί τις αμφιβολίες μας. Γεγονός είναι πάντα ότι έχετε ένα φορολογικό καθεστώς ιδιαίτερα περιορισμένο. 10% στις εταιρείε, πάρα πολύ για νεόδοροι, κάνετε εκπτώσεις ή μάλλον φορολογικές ελαφρύνσεις για ε, την ε, ε, πνευματική διοκτησία, για τις ενδομιλικές συναλλαγές και μάλιστα το διαφημίζετε. Πηγαίνετε στην Ισπανία και κάνετε διαφήμιση και εξηγείτε ότι ελάτε στην Ανδώρα παρακαλώ, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Γιατί έχουμε φορολογικές ελαφρύσεις. 900 επιχειρήσεις από το 2012 έχουν φύγει από την Ισπανία και πάνε στην Ανδώρα. Ε, και θυμίζω ότι ε, ε, έχετε μόνο 70.000 κατοίκους, 900 επαναλαμβάνω. Και πιστεύετε ότι μετακομίζουν οι εταιρείε μόνο για φορολογικούς λόγους ή υπάρχει και οικονομική δραστηριότητα υποκείμενη. Και μια δεύτερη ερώτηση θέλω να μου απαντήσετε συγκεκριμένα. Συμφωνείτε με την Επιτροπή μας ότι τα κέρδη θα πρέπει να φορολογούνται εκεί που παράγονται και όχι εκεί που εγγράφονται λογιστικά. Και θεωρείτε ότι είναι σωστό αυτό ως άποψη της Επιτροπής μας. Υπάρχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ανδώρα και δραστηριοποιούνται παντού στην Ένωση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά συμβαίνει το εξή. Στην Ισπανία υπάρχουν εταιρείε που κάνουν φορολογική δήλωση. Εταιρείε, έτσι. Ε, φυσικά και νομικά πρόσωπα με, ε, εθνικότητα Ανδόρας. Και κάνουν κάθε τρίμηνο ε, μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ή κάποιες θετικές και μετά ποτέ δεν πληρώνουν. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία σύμβαση για αμοιβαία συνδρομή σε θέμα εκτέλεσης αποφάσεων. Ε, σκέφτεστε να κάνετε καμιά τέτοια κίνηση, να υπογράψετε κάτι με την Ισπανία για την φόρου, ναι ή ου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας τώρα. Θα ήθελα να αρχίσουμε με την Ανδώρα θα επανέλθουμε σε αυτό ε, για τα ερωτήματα των που πρέπει να αναχωρήσει και εξάλλου ε, σχετίζεται και με άλλα γενική φύσεως ερωτήματα. Um, thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με τη σειρά που επιθυμώ. Ίσως μπορώ να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Καλώς. Καλώς. Μπορώ να μιλήσω ισπανικά. Ορίστε. Μα χρησιμοποιείτε όλε τι επίσημε γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Επειδή επέβαλε την ερώτηση στα ισπανικά. Θα απαντήσω ισπανικά. Ε, Σε σχέση με την τελευταία ερώτηση, που είναι η γειτονική μα χώρα και μία από τι χώρε με τι οποίε έχουμε τι περισσότερε σχέσει και στη συνέχεια θα απαντήσω στις ερωτήσεις για το ποιες είναι οι χώρες με τις οποίες έχουμε περισσότερες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές σχέσεις. Η Ισπανία είναι μία από τις σημαντικές μας γειτονικές χώρες και εταίρους και επαναλαμβάνω και πάλι ότι ε, φορολογικός παράδεισος δεν είμαστε. Κάναμε πολλές αλλαγές, ε, παρακολουθήσαμε και σας είπα προηγουμένως από το 2009 μέχρι σήμερα όχι μόνο ανοίξαμε την οικονομία μας αλλά Έχουμε επιβάλει όλη τη φορολογία ε, που οφείλαμε και είναι μεγάλο βήμα αυτό μέσα σε τέσσερα χρόνια. Επίσης, ακολουθούμε όλους τους κανόνες της διαφάνειας και τώρα ε, είμαστε στο θέμα του BEPS, της ομάδας εργασίας, συνεργαζόμαστε. Σε ό,τι αφορά το θέμα τώρα της επιβολής φορών, η φορολογική μας βάση είναι πολύ απλή, διότι είναι 10% ε, ενιαίος φορολογικός συνδελεστής. Ε, αλλά εμπνεώμεθα εμείς από το φόρο που επιβάλλουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα και διεθνώς. Υπάρχει αυτό. Όπως σας είπα, βέβαια πάντα εγγραφόμαστε ε, στη διαφάνεια, στις βέλτιστες πρακτικές και ό,τι άλλο ισχύει. Βεβαίω όλες τις ομάδες εργασίας συμμετέχουμε, αναθεωρούμε ό,τι χρειάζεται για να ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και πρέπει να σας πω ότι όταν κάναμε τις συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, ε, συζητούμε αυτά τα θέματα και δεν υπήρχε ποτέ κανένα πρόβλημα για να υπογράψουμε αυτές τις συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολόγησης. Άρα, το Φεβρουάριο 26 του σε ετέθησε ισχύ η συμφωνία με την Ισπανία και τώρα διαπραγματευόμαστε να δούμε για το ποιο είναι ο και η φορολογική βάση και η κατάσταση σε ε, διάφορες καταστάσεις και έχουμε και ρήτρε κατά των καταχρήσεων. Δηλαδή, αν έρχεται κάποιος να εγκατασταθεί στην Ανδώρα είναι για να ασκήσει εκεί μια δραστηριότητα, χωρίς όμως αυτό να είναι εις βάρος κάποιου άλλου. Είναι, είναι ε, εικονική πραγματικότητα ή να το εκμεταλλευτεί ε, για να μην ε, πληρώνει φόρους πουθενά. Οπότε, σε όλα αυτά και πέρα από τις συμφωνίες γιατί είναι πολύ ε, πρόσφατες και στο BEPS ε, συζητούμε για όλες ε, τις ρήτρε κατά των καταχρήσεων κτλ. Και θα πρέπει να πούμε ότι σε όλες αυτές τις ομάδες εργασίας των ΠΕΠΣ που συμμετέχουμε από την αρχή έχουμε και πολυμερείς διαπραγματεύσεις, λαμβάνουμε υπόψη όλες τις δράσεις. Είμαστε μικρή χώρα και προσπαθούμε ε, όσο γίνεται συμμετέχουμε σε περισσότερα φόρα, παρακολουθούμε τα πάντα. Τώρα αν υπάρχουν κάποια σημεία που χωρούν βελτίωση, είμαι η πρώτη που θα πω ότι ναι, ως εκπρόσωπος της Ανδόρα παντού θα ρωτήσω τι χρειάζεται για να ε, προσαρμοζόμαστε πάντα στο διεθνές ε, στερέωμα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σεβόμαστε και να συμμορφούμαστε προ τι διεθνείς προδιαγραφέ και δεν ξέρω να απαντά λίγο στην ερώτησή σας αυτό. Σας ευχαριστώ για τις άλλες ερωτήσεις που ετέθησαν, κυρίως από τον εισηγητή, τον κύριο Έγκελ. Πολύ γρήγορα παρακαλώ. Ε, Όσον αφορά τον ΩΣΑ και τη διαφορά με τη συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπογράψαμε το 2005 και αυτή που έχουμε τώρα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη διαφορά, διότι αν ρίξετε μια ματιά θα δείτε ότι είναι η ίδια με αυτή του ΟΣΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών, όλων των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται για τον ΟΣΑ. Επί της ιδίας βάσεως θα δίνουν πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήρη ανταλλαγή πληροφοριών, όπως θα κάνουμε και για τις άλλες χώρες. Υπογράψαμε ήδη πολυμερή συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές, ετοιμάζουμε όλη την ομοθέσια, το λογισμικό κλπ. ούτω ώστε του χρόνου να γίνει η δοκιμή, να ξέρουμε ότι λειτουργεί το σύστημα. Η αλλαγή είναι πολύ μεγάλη, διότι θα γίνεται πλήρη ανταλλαγή πληροφοριών. Ερώτηση του Πρόεδρου. Η έκθεση αναχώρα θα αποκαλύπτει τα στοιχεία αυτών. Είναι κάτι που μελετούμε η απάντηση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και θέματα. Αν όλοι συμμετέχουν, γιατί να μην συμμετάσχει και δώρα, Θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε εκεί, παρακολουθούμε τι γίνεται, τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο, αναλύουμε τον αντίκτυπο και προσπαθούμε να δούμε πως θα κινηθούμε. Όπω με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν εκείνοι που το εφαρμόζουν πιο έγκαιρα και άλλοι που θα το εφαρμόσουν το σύστημα το 2018 πρέπει να δούμε ποιος είναι ο δικός χάρτης, ποια είναι η πορεία και πότε θα ήταν δυνατόν να τα εφαρμόσουμε αυτά. Ε, the... Όσον αφορά την μεταφορά της τιμολόγησης, το φορολογικό πλαίσιο είναι νέο, νεότατο. Έχουμε αρμόδιο φορέα που ξεκίνησε τις εργασίες πέρσι. Πολύ καινούριο φορέας. Θα αναπτύσσουμε όλα αυτά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο. Θα δούμε τι χρειάζεται για να ανταποκριθούμε σε απαιτήσει Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Το φορολογικό σύστημα είναι πολύ απλό αυτό που έχουμε τώρα. Πολύ γραμμικό. Έχουμε ήδη ετοιμάσει ομάδες εποπτείας. Θέλουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστούν οι λεπτομέρειες για τα φορολογικά. Πώς μπορούν να εφαρμοστούν, αν υπάρχει σωστή προσέγγιση ή όχι, αν συνομορφωνόμαστε με τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις διεθνείς προδιαγραφές. Οπότε έχουμε δρομολογήσει την ανάλυση αυτών. Μέχρι τώρα έπρεπε να οργανώσουμε το σύστημα. Είναι πολύ δύσκολο για μια μικρή χώρα να ε, κανονίσει τα των φόρων και των φορολογικών φορέων, αρμοδίων φορέων. Θέλουμε να μελετήσουμε τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο και να αναρμονιστούμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκτός συντονισμού. Θέλουμε να συντονιστούμε με τις άλλες χώρες. Κύριε Φυπουργέ, ναι, μιλάω κάτι γερμανικούλια, αλλά καλύτερα να ακούσω τίποτα άλλο. Δεν είναι πολύ ικανοποιητικό αυτό που μας απαντάτε ότι το ελέγχετε και το εξετάζετε αυτό τον καιρό. Εντάξει, μπορώ να καταλάβω ότι εξετάζετε κάποια πράγματα, αλλά μήπως να είστε λίγο πιο ενημερωτικοί και να μας πείτε τι επιφυλάξεις έχετε ε, σε σχέση με ρυθμίσεις που προτείνονται, τι θα σας εμπόδιζε. Ξέρω ότι όλα αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά μήπως να μπείτε λίγο περισσότερο στην ουσία και να μην το διεκπαιρεώνετε έτσι και, και κάπως ε, ε μας λέτε ότι το εξετάζετε αυτό καιρό χωρίς να απαντάτε. Ίσως θα σας βοηθούσε να σας πω ότι για το φόρο των επιχειρήσεων θέλετε να γνωρίζετε πώς λειτουργεί. Αυτό θέλετε. 10% φορολογικό συντηρητής Έχετε μειώσεις αν δημιουργείτε νέες θέσεις εργασίας. Ή μια νέα επιχείρηση. Αν πληρώνετε τοπικό φόρο. Για την τοπική αυτοδίκηση. Για να αποφευθεί διπλή φορολόγηση υπάρχουν κάποιες ελαφρύνσεις. Και κάποιες ειδικές ελαφρύνσεις. Σύμφωνα όμως με ειδικά καθεστώτα που αφορούν το διεθνές εμπόριο. Διαχείριση διαφόρων οικονομικών επενδύσεων εντός ομίλου και με κάποιες επενδύσεις στο εξωτερικό, κάποιες συμμετοχές στο εξωτερικό. Πρέπει να γίνει σωστή ανάλυση. Να δούμε αν επιτρέπεται αυτή η κίνηση ή όχι. Δεν είναι κάτι αυτόματο. Κατά περίπτωση γίνεται η ανάλυση για τις ελαφρύνσεις. το, ονομαστικό το ονομαστικός φορολογικός συντελεστής είναι 10%. Σχεδόν πάντα έχουμε 10%. Και έχουμε μόνο τις ελαφρύνσεις που ανέφερα. Αν δημιουργείται νέους τομείς, νέες θέσεις απασχόλησης, αν αυξάνεται η επιχειρηματικότητα στη χώρα, υπάρχουν ελαφρύνσεις. Αλλιώς όλοι πληρώνουν αυτό το φόρο 10% δεν μεταβάλλεται κατά πολύ. Το θεωρητικό φορολογητέο ποσό με αυτό που υπάρχει πραγματικά είναι το, σχεδόν το ίδιο. Όταν λέω αναλύουμε, δεν αναλύουμε το δημοσιονομικό, το φορολογικό μας πλαίσιο. Αυτό το αναλύσαμε πριν εφαρμοστεί. Τι λέω τώρα. Με τα BEPS και με τις συμβάσεις περί αποφυγής της φορολόγησης γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κανόνες κατά των καταχρήσεων. Και κατά σύμβαση κάνουμε αναλύσεις για να δούμε ποιος μπορεί να είναι αντίκτυπος να έχουμε διαφορετική φορολόγηση. Στην πολυμερή ομάδα για τα BEPS συμμετέχουμε και βλέπουμε ότι όλοι αναλύουν εκεί, όχι μόνο εμείς. Θέλουν να δούνε ποιος είναι αντίχτυπος των νέων δράσεων. Τι θέλω να πω με όλα αυτά αναλύουμε όλα τα τεκτενόμενα. Διότι πρέπει να αφιγραμμιστούμε. Και αν υπάρχει κάτι καινούριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούμε. Γι' αυτά υπογράφουμε συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ΟΣΑ, το ίδιο με τις ΗΠΑ, με όλους. Πρέπει όμως να έχουμε έναν οδικό χάρτη, ένα προσανατολισμό, να είμαστε σίγουροι ότι ό,τι κάνουμε ευθυγραμμίζεται με όλα αυτά και να έχουμε τον κατάλληλο χρόνο να εξετάσουμε τα πάντα. Ευχαριστώ, λέει Η κυρία ο Πέτερ έχει το λόγο. Δεν απαντήσατε. Δεν απαντήσατε την ερώτηση Γιατί είναι αυτό με την ανταλλαγή πληροφοριών ε, για τα tax rulings. Υπάρχουν τέτοιε φορολογικές αποφάσει. στην Ανδόρα. Γιατί αυτό εξετάζουμε εμείς και αν γίνει αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετέχει ενδόρα σε αυτό το σύστημα. Madame. Ορίστε. Δείχνουμε ότι συμμετέχουμε σε όλα τα νέα μέτρα, σε όλα όσα εξελίσσονται. Αν υπάρχουν νέοι κανόνες, θα δούμε τι συμβαίνει. Θα δούμε πώς μπορούμε να τι εφαρμόσουμε. Αν δεν θέλαμε να ακολουθήσουμε, να συμμορφωθούμε με όλου του διεθνεί κανόνε και του ευρωπαϊκού και του άλλου κανόνε, δεν θα ήμασταν εδώ. Βεβαίω αυτό θέλουμε. Η απάντηση λοιπόν είναι ναι, λέει ο Πρόεδρο. Στα πάντα ναι. Σε όλα ναι. Σε όλα αυτά που πρέπει. Πρέπει να δούμε τι κατευθύνσει στον οδικό χάρτη. Να γραφεί τα πρακτικά παρακαλώ αυτό το ναι σε όλα. Μάλιστα, η κυρία Γκέιλ. <coughs> Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελπίζω να έχω καταγράψει όλες τις υποβληθείς ερωτήσεις στις αναχώρα εκθέσεις. Ναι, υποστηρίζουμε τα BEPS όσα εν γέννη. Ναι, έχουμε υπογράψει την πολυμερή συμφωνία της αρχές για αναχώρα υποβολή εκθέσεων, κάτι που έχει ετοιμαστεί από τον ΩΣΑ. Θα εφαρμοστεί αυτό σύμφωνα με τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας στην αρχή της κυβέρνηση αρχές Μαρτίου, όπως ανακοινώθηκε στον τύπο, ήδη ξεκίνησε την υλοποίηση ενός πρώτου νομοθετικού πακέτου. Θα υποβληθεί αυτό το πακέτο μάλλον για διαβούλευση. Για την εφαρμογή των BEPS. Πρώτα πρέπει να θεσπιστεί κατάλληλη νομοθεσία για την υποβολή ε, εκθέσεων αναχώρα σύμφωνα με τι απαιτήσει όσα άλλο μέτρο που θα αφορά τη σταδιακή εξάλληψη του καθεστώτος με τα διάφορα τετραγωνίδια που χρησιμοποιούσαμε εντός της μεταβατικής περίοδου μέχρι το τέλος του 2020 με άλλα λόγια. Θέλουμε στο νόμο μας για τη φορολογία να έχουμε σαφή ορισμό του ruling, της αποφάσεως φορολογικής και ορισμός αυτός μετά θα χρησιμοποιείται για τη σωστή ανταλλαγή τέτοιων αποφάσεων, rulings. Έχουμε σχεδιάσει επίσης και κάτι άλλο. να θεσπιστεί και εθνική νομοθεσία την ε, τιμολόγηση των διαφόρων μεταφορών και τιμολόγηση της, των μετατοπίσεων που θα πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το θέμα σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΣΑ. Τώρα το άλλο ερώτημα που αφορά την υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Αν πρέπει να δημοσιοποιούνται ή όχι τα στοιχεία. Πιστεύουμε ότι μέχρι τώρα τίναμε να ακολουθούμε τα συμπεφωνημένα σε διεθνές επίπεδο, τις σχετικές προδιαγραφές του ΩΣΑ Αυτά θα εφαρμόζαμε ως προσέγγιση. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες κατά πόσο η δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του επιχειρηματικού απορρίτου αν οδηγεί σε προστιθέμενη αξία. Αν βέβαια θεσπιστούν διεθνείς προδιαγραφές που προβλέπουν κάτι τέτοιο, ότι πρέπει να δημοσιοποιούνται δηλαδή αυτές οι πληροφορίες και να ανταλλάσσονται, τότε ασφαλώς θα προσαρμοστούμε δεόντως. Όπως και κάθε άλλη χώρα. Υπήρξε άλλη ερώτηση όσον αφορά τα ιδρύματα, καταπιστεύματα, επιχειρήσεις, κεντρικά μητρώα πραγματικής ιδιοκτησίας και τις συναφείς πληροφορίες. Στην πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης του Global Forum είδατε ότι έγινε αξιολόγηση και ότι οι πληροφορίες περί ιδιοκτησίας όσον αφορά τις εταιρείες ιδρύματα, καταπιστεύματα και άλλες οντότητες είναι στοιχεία διαθέσιμα στο Λίχτενστάιν. Όχι δημοσίως όμως, δημοσιοποιούνται αυτά τα στοιχεία κανονικά. Είναι διαθέσιμα όμως. Αυτό είναι το σημαντικό. Όσον αφορά την ανάγκη των αρχών να έχουν πρόσβαση σε αυτού του είδους τις πληροφορίες που εν γέννη βρίσκονται εντός των αρχείων των εταιριών και των παρόχων υπηρεσιών είναι πολύ ανεπτυγμένο το σύστημα, επί σειρά ετών ανεπτύσσετο και η εμπειρία για την ανταλλαγή πληροφοριών καταδεικνύει ότι μέχρι τώρα δεν υπήρξε περίπτωση όπου δεν μπορούσαμε να βρούμε ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης πίσω από κάποιο ίδρυμα ή κάποιο καταπίστευμα ή οποιονδήποτε άλλο φορέα. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε αποδεδειγμένο ιστορικό όσον αφορά την διαθεσιμότητα του νόμιμου πραγματικού ιδιοκτήτου και των σχετικών πληροφοριών. Πέραν αυτού, όχι μόνο με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν ετήματος αλλά με τη μελλοντική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα παραλαμβάνετε όλα τα σχετικά κείμενα και πληροφορίες για αυτούς τους πραγματικούς ιδιοκτήτες αυτομάτως βάσει ευρυτέρου τώρα ορισμού του ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Μετά υπήρχε άλλη ερώτηση. Εάν την κατανόησα, κατανόησα σωστά στον αφορά την πρακτική που ακολουθείτε για η ειδική φορολογική δικαιοδοσία, πόσο σημαντική θα ήταν αυτή για τη χώρα και ποιες προνομιούχες σχέσεις έχουμε με τους γείτονές μας, αν υπάρχουν τέτοιες προνομιακές σχέσεις και από πού προέρχονται, από ποιες χώρες προέρχονται οι επενδυτές μας. Εν γέννη, δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά την προέλευση των επενδυτών στις διάφορες επιχειρήσεις. Όμως, εν γέννη, μπορώ να σας πω ότι έχουμε πολύ στενές οικονομικές σχέσεις βεβαίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός του οικονομικού χώρου, όχι μόνο στον τομέα τον οικονομικό, το χρηματοδοτικό και στο βιομηχανικό όμως. Όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτής, αλλά και με τις Ηνωμένε Πολιτείες και με ασιατικές χώρες και με χώρες της Αμερικανικής Υπήρου και της Νοτιού Αμερικής συμπεριλαμβάνονται. Και Ελβετία λέει ο Πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήρθαν παρόλο. Βέβαια, βέβαια. Δεν είμαι σίγουρη ακριβώς ποιος ήταν ο στόχος ερωτήσεως. Ήθελα να πω ότι κατά την άποψή μου δεν είναι τόσο σημαντικό να δούμε ποιες ακριβώς δραστηριότητε λαμβάνουν χώρα σε μία χώρα. Αλλά κατά πόσο αυτές οι δραστηριότητες είναι νόμιμες και αν συμμορφώνονται με διεθνείς προϋποθέσεις και απαιτήσει και ευρωπαϊκές, αν τεκμηριώνονται σωστά αυτές οι δραστηριότητες. Και αν χρειάζεται για τον καθορισμό των φόρων να γίνεται σωστή ανταλλαγή πληροφοριών. Ακριβώς αυτό ισχύει για το Λίχτενστάιν. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι ανταλλαγές πληροφοριών. Επ' αυτού ο Φρανκ Έγγελ θέλει κάποια διευκρίνηση, να διευκρινίσει την ερώτησή του μάλλον. Αν επιτρέπετε ο Φρανκ. Αγαπητή κυρία Κάι, θα τα πω γερμανικά για να καταλαβαίνόμαστε καλύτερα. Δεν ε, σας προσάπτω ότι κάνετε κάτι κακό και ε, σας ρώτησα φιλικά τι κάνετε και ε, αν θέλετε να μας πείτε αν έχετε tax rulings. Μέχρι τώρα δεν έχετε απαντήσει. Είναι θεμητή ερώτηση. Κανονικά ε, θα πρέπει να έχω τη δυνατότητα και καλοπροαίρετα να την κάνω. Αν ήμουν λιγότερο καλό, θα ρωτούσα γιατί χρειάζεται στο Liechtenstein ένα ίδρυμα σε σχέση με την ελβετική δικαιοδοσία για να προσπαθήσει κανείς να αποφύγει τη φορολόγηση. Δεν το είπα έτσι γιατί ήθελα να είμαι καλός. Τώρα μάλλον θα αγριέψω λίγο. Τότε να απαντήσω και εγώ γερμανικά για να με καταλάβετε καλύτερα. Ja, es gibt... Ε, ναι, υπάρχουν ε, tax rulings στο Liechtenstein, μάλιστα. Είπα εισαγωγικά ότι αυτές οι συμφωνίες οι φορολογικές ελέγχθησαν από την εποπτική αρχή της ΕΖΕΣ που είναι το αντίστοιχο ομόλογος ας πούμε το όργανο αυτό στην, ε, ε, στον ΕΟΧ της, στην ΕΖΕΣ συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρακολουθεί την εσωτερική αγορά και κοιτάει τι γίνεται με τις κρατικές ανισχύσεις και εποπτεύει και παρακολουθεί. Οι φορολογικές συμφωνίες αυτές, τα tax rulings που που ελέγχθησαν μάλλον και που δώσαμε στοιχεία στην ΕΖΕΣ όπως κάνουν κατά τα άλλα και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έλεγξα λοιπόν αυτά τα στοιχεία και κατέληξε η αρμόδια αρχή ότι οι δικές μας πρακτικές να κάνουμε τέτοιες φορολογικές συμφωνίες tax rulings ε, συνάδουν με τους ευρωπαϊκούς κανόνες που ισχύουν και εφαρμόζονται και ιδιαίτερα με τις διατάξεις για την αποφυγή κρατικών ενισχύσεων. Έχει εδώ σημασία να πούμε ότι σε εμά οι φορολογικές συμφωνίες, tax rulings, σε καμία περίπτωση δεν έχουν στόχο να μειώσουν το φόρο, αλλά αποκλειστικά και μόνο να παρέχουν ασφάλεια δικαίου για το πώς θα φορολογούνται οι επιχειρήσεις βάσει του ισχύοντος δικαίου για ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο που και πολύ συγκεκριμένα πρέπει να υλοποιείται. Σε περίπτωση που δεν γίνεται κάτι τέτοιο, τότε είναι άκυρη αυτή η συμφωνία. Ελπίζω να απάντησε στην ερώτησή σας. Αν έχουμε φορολογικές συμφωνίες τύπου tax rulings ή όχι. Για την νομιμοποίηση. κάποιων δυνατοτήτων που έχουν οι εταιρείε ε, που τις χρησιμοποιούν ή όχι. Ένα από τα βασικά θεμέλια της Ευρώπης είναι η εσωτερική αγορά. Και η ευκαιρία επενδύσεων στην ενιαία αγορά, όχι μόνο στην πατρίδα του καθένα. Αυτό είναι από τα ίδια τα θεμέλια ε, τη εσωτερική αγορά και του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Εμεί το τηρούμε αυτό και συμμετέχουμε. επίση τηρούμε και όλου του κανόνε που συνδέονται με αυτό. Τώρα, όταν πρόκειται για ε, φορολογική ε, δημιουργικότητα ε, θα πρέπει να δούμε τα νέα στάνταρ και τις προγραφές του ΩΣΑ και το σχέδιο ΠΕΠΣ για τη διάβρωση της βάσης και τη μεταφορά των κερδών. Το κάνουμε και για τα rulings αλλά και με κάποιες επιμέρους ε, εκάστοτε προσαρμογές στο φορολογικό μας δίκαιο. Εδώ ίσως θα πρέπει να αναφέρουμε ιδιαίτερα ότι η γενική απαλλαγή μερισμάτων ε, και ε, εισοδημάτων από μερίσματα θα εγκαταληφθεί. Όπως επίσης και ε, άλλωστε αυτό αναφέρεται στην αντίστοιχη οδηγία για τις μετρικές και θηγατρικές εταιρείες. Ακριβώ αφενός για να αποφευθεί διπλή φορολόγηση και αφετέρου για να αποφευθεί στο μέλλον ενδεχομένως βρυδική μορφή οντότητων, οντότητες. Αυτά μπορώ να σας πω σήμερα. Δεν είμαι σίγουρη, μήπως ξέχασα να απαντήσω ε, μία ερώτηση. Α, ναι. Ρωτήσατε πώς ε, αξιολογούμε την προηγούμενη συμφωνία για την ε, φορολόγηση των, καταθέσεων, των αποταμιεύσεων, των καταθέσεων και κατά πόσο κρίνουμε θα είναι αποτελεσματικότερη η τωρινή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω όλοι γνωρίζουμε πως οι συμφωνίες φορολόγησης καταθέσεων και η προηγούμενη ενισχύ για τη φορολόγησή τους είχαν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Ε, ως εκ τούτου ήταν περιορισμένη και αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι συμφωνούσαμε από αυτού. Εντός του πεδίου εφαρμογής είτε είχαμε ε, εισπράξει τους φόρους και τους μεταφέρει στα κράτη-μέλη ή σε μεγαλύτερο ακόμη βαθμό είχαμε ανταλλάξει σχετικές πληροφορίες. Φυσικά θα είναι πάρα πολύ αποτελεσματικότερη η νέα συμφωνία διότι είναι ευρύτερη και καλύπτει περισσότερες κατηγορίες ε, εσόδων Φυσικά και με τη θέσπιση αυτόματης ανταλλαγής ε, πληροφοριών έχουμε ένα γενικό και κοινό πρότυπο που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά όμως και με τους εταίρους μας ε, δυνάτων ε, ενισχύσεις συνθήκων. Πίτερ, θέλετε να επανέλθετε για την ερώτηση του Μπέντ. Μόνο για να διευκρινίσουμε κάτι. Είπατε εισαγωγικά ότι ότι εφαρμόζεται τη ρύθμιση των χρηματαγορών. Δηλαδή αν έχουμε αυτόματη αταλλαγή προφοριών για τα tax rulings θα το εφαρμόσετε και την κοινή ενοποιημένη βάση για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων ε, και ένα μητρό δημόσιο ε, μάλλον ε, αναφορά αναχώρα αν είναι δημόσια αλλιώς θα συμμετέχετε σε αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ για τη συμπληρωματική ερώτηση. Κοιτάξτε, θα πρέπει να σα υπενθυμίσω εδώ ότι το Λίχτενστάιν δεν είναι κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά ότι εφαρμόζεται την νομοθεσία για τις χρηματαγορές. Ναι, για τις χρηματαγορές την νομοθεσία την εφαρμόζουμε βεβαίως. Αλλά τη φορολογική νομοθεσία, ε, υπάρχει ένα φορολογικό κεκτημένο ε, στην Ένωση και δεν είναι τμήμα τη Συμφωνία του ΕΟΧ αυτή. Και αυτές οι διατάξεις δεν καλύπτονται από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. Και μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έχει κάνει καμία ανοίξη ή καμία πρόταση να διαθετήσουμε ε, και άλλα τμήματα του φορολογικού της κεκτημένου, είτε προτάσεις να αρχίσουν διαπραγματεύσεις και τέτοια πράγματα. Ούτε για την ανταλλαγή ε, ε, πληροφοριών για τα tax rulings, ούτε για τη δημιουργία μιας κοινή φορολογικής βάσης για μια κοινή ενοποιημένη φορολογικής βάσης. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω, δυσκολεύομαι γιατί μέχρι τώρα δεν ήταν για μας ζήτημα στις σχέσεις μας ε, με, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η απάντηση είναι αρνητική, μάλιστα. Νάιν δηλαδή. Ο Μπεντ Λούκε, ναι, στην ίδια κατεύθυνση να πω κάτι, γιατί δεν απαντήθηκε, νομίζω, δεν μας απαντήσατε. Σα ρώτησα αν πιστεύετε ότι η εισαγωγή μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε αρνητικέ συνέπειε ε, για τα φορολογικά έσοδα του Λίχτενστάιν αν γίνει αυτό προς αποφυγή διπλής φορολόγηση. Και βεβαίως ε, δεν είστε υποχρεωμένοι να υιοθετήσετε το φορολογικό κεκτημένο, αλλά τίποτα δεν σας εμποδίζει να το κάνετε εθελοντικά. Θα κινούσετε μια τέτοια πρωτοβουλία. Um, wie Aus... Όπως σας είπα, οι επιπτώσεις μια κοινή ε, ε, ή μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων είναι κάτι που εμείς ακόμα δεν έχουμε αναλύσει. Για να μπορώ να σας δώσω μια αξιόπιστη απάντηση. Μια κοινή φορολογική βάση μπορεί να έχει κάποια πλέον εκτίματα. Τώρα μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση ε, με αναδιανομή ε, των φορολογικών εσόδων μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να έχει κάποιες επιπτώσεις ενδεχομένως. Για εκείνους που δεν είναι τμήμα του συστήματος κυρίως. Τώρα, ε, σε ποιο βαθμό και πόσο σημαντική θα είναι αυτή η επίπτωση είναι δύσκολο μέχρι στιγμής να το αξιολογήσουμε. Αν με ρωτάτε αν θα προσχωρήσουμε σε αυτές τις νέες ρυθμίσεις, Μέχρι τώρα, σχέσεις Λίχτενστάιν και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, ε, δράζονται σε, πάρα πολύ σαφείς συμβατικές υποχρεώσεις. Οι συνθήκες έχουν και πολλές υποχρεώσεις αλλά και, πολλά, και κάποια δικαιώματα. Άρα, αν κάποιος διευρύνει τις υποχρεώσεις που οφείλουμε να εφαρμόσουμε, τότε φαντάζομαι το Λίχτενστάιν θα υιοθετήσει τη θέση που λέει ότι να ε, διευρυνθούν και τα δικαιώματα που μπορεί κανείς να αποκομίσει από μια τέτοια συμφωνία για να υπάρχει μια εξισορρόπηση κάπου και να μπορεί να εφαρμόζεται και το όλο σύστημα. Για παράδειγμα, αυτό θα σήμαινε ότι ορισμένες οδηγίες για την αποφυγή διπλής φορολόγησης που αυτή τη στιγμή δεν έχουν επεκταθεί στο Λίχτενστάιν, όπως είναι η οδηγία για τη μετρική θηγατρική εταιρεία ή, ή για τη, τους τόκους, θα πρέπει να είναι τμήμα της συμφωνίας αυτής. Και ούτε θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε πράγμα που σήμερα είναι ήδη απαράδεκτο το Λίχτενστάιν να παραμένει σε κάποιες μαύρες λίστες ορισμένων κρατών μελών ή να θεωρείται ε, αρνητικό και να ε, υφίσταται ε, αρνητικές διακρίσεις. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο ήδη από τώρα γιατί υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Παρ' όλα αυτά, πολλά και ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διστάζουν να αφαιρέσουν το Λίχτενστάιν από τη μαύρη λίστα. ή διάφορε μαύρες λίστες που διατηρούν για λόγους έλλειψης πληροφοριών με τις εν λόγω χώρες. Κατά τα άλλα υπάρχει και διακριτική μεταρρύθμιση, μεταχείριση σε μαύρες λίστες που μας κατατάσσουν σε επιζήμια φορολογικά συστήματα ή ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις ε, ως προς το φορολογικό συντελεστή. Σε αυτό το γενικό πλαίσιο λοιπόν θα πρέπει να το κοιτάξουμε σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο γιατί κατά την άποψή μας αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τόσο πολύ να επιβληθούν μονομερώς ορισμένες ε, ρυθμίσεις που αποφασίζει το ιστορικό η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ δε περισσότερο που το Liechtenstein είναι τμήμα της ευρωπαϊκής αγοράς και δεν είναι μια τυχαία οποιαδήποτε τρίτη χώρα, όπως σας είπα εισαγωγικά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κοφότ θέλει να κάνει μια επερώτηση. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ. Επερώτηση. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο τα καταπιστεύματα και την, ε, το καθεστώς ιδιοκτησίας τέτοιων ιδρυμάτων γιατί δεν μπορείτε να τα κοινοποιήσετε. Και δεύτερον, για τις ε, εταιρείε ε, δημοσίου συμφέροντος, αν κατάλαβα καλά την απάντησή σας, πληρείτε τις απαιτήσει του ΩΣΑ, ναι μεν, όμως δεν έχετε επίσημο μητρό για το καθεστώς ιδιοκτησίας προ το παρόν, για αυτές τις επιχειρήσεις ούτε και ε, δημοσιεύετε λογαριασμούς για τις ΔΕΚΟ. Μπορείτε να μας ε, ενημερώσετε γιατί εγώ κάθε άλλο παρά διαφανή σας βρίσκω. Αν μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Απάντηση. Φυσικά έχουμε μητρό επιχειρήσεων και θα έχετε και πρόσβαση. Αυτό που δεν έχουμε είναι δημόσιο μητρό ιδρυμάτων και άλλων δοτήτων. Όμως, όταν ιδρύονται αυτές οι οντότητες, παρόλα αυτά πρέπει να καταχωρίζονται στην, στο μητρό. Τι σημαίνει αυτό. Η σύσταση των ιδρυμάτων εποπτεύεται εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες ως προς το καθεστώς ιδιοκτησίας φυλάσσονται παρότι όχι σε δημόσιο μητρέο. Για τις ε, εταιρείε ε, που είναι συγμένες στο χρηματιστήριο εξυπακούεται ότι πληρούμε όλες τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Δεν είμαι σίγουρη για τις πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας των εταιριών, κυρίως για τις ανώνυμες εταιρείες, αν η διαφάνεια ε, ε, για το κοινό μπορεί να εκλειφθεί ως ε, παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό πρότυπο. Εν τη περιπτώσει σημαίνει η διαφάνεια πως συντρέχει κάποιος λόγος. Ε, χάρη, ε, νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων, οικονομικά εγκλήματα, φορολογικές ε, πληροφορίες. Έτσι το καθεστώς ιδιοκτησίας όλων των εταιριών ε, trust, καταπιστευμάτων και foundation συνδρυμάτων συνιστούν πληροφορίες που απαιτούνται να κοινοποιηθούν αλλά αυτό δεν ισοδυναμεί με μια πάγια υποχρέωση ε, δημόσιας πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες δεν διαπιστώνω δε μία προστιθέμενη αξία σε μια τέτοια απέτηση, ούτε εξάλλου ε, και σε σχέση με την διαπίστωση φορολογικής συμβατότητας ε, πρόληψης νομοποίησης παρανόμων εισόδων, ε, εσόδων συγγνώμη, ή χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων. Γι' αυτό το λόγο φυσικά προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο σύστημα και έχουμε θεσπίσει ένα σύστημα ως προς το καθεστώς ιδιοκτησίας και νομικό καθεστώς αυτών των εταιριών. Είναι πα... πάγια προσβάσιμες αυτές οι πληροφορίες. Όμως ε, δεν εξασφαλίζεται απαραίτητα δημόσια πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. ευχαριστούμε. Στρέφομαι προς το Μονακό. Υπουργέ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τις ερωτήσεις που αφορούν όλος ιδιαίτερος στο πριγκιπάτο διότι έχω την εντύπωση ότι απέφθηναν οι βουλευτές ε, μάλλον τα περισσότερα ερωτήματα στους ε, υπόλοιπους συμμετέχοντες. Λοιπόν, εφαρμογή των, ε, της 2005 και απολογισμός της εφαρμογής προς υπογράφω αυτά που είπε η πρόσωπος του Λιχτενστάιν. Οι διατάξεις ήταν εκφύσεως μεταβατικές με περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Παρόλα αυτά επέτρεψαν στο πριγκιπάτο να συλλέξει ποσά που με μετέφερε στα κράτη-μέλη εδώ και μία δεκαετία και δεν είναι διόλου αυτά τα ποσά. Όμως, να τονίσουμε επίσης ε, την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος βάσει συμφωνίας με τον ΩΣΑ από το 2009 και μετά. 30 περίπου συμφωνίες έχουμε υπογράψει και ε, ως επιτοπλίστων ισχύουν σήμερα και ανταλλάσσουμε πληροφορίες κατόπιν αιτήματος με πολλές χώρες Έχουμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ε, και τα αποτελέσματα σε διάφορα παγκόσμια φόρα που ε, έλαβαν χώρα μας έδωσαν πολύ θετικές αξιολογήσεις για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, ε, την ΜΑΚ, την MCA έχουμε υπογράψει. Ακολουθούμε αυτό το παγκόσμιο κίνημα. Φυσικά η κάνουμε τον απολυσμό των προηγουμένων συμφωνιών, αλλά κυρίω εντασσόμεθα σε αυτήν τη νέα δυναμική των νέων παγκοσμίων συμφωνιών. Θα ήθελα για τα υπόλοιπα ερωτήματα να δώσω ένα είδος απάντηση και ενδεχομένω να κάνω και διευκρινή συνέχεια. Ο κύριος Αντώνη Ελκέν που είναι ο διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών θα ήθελα να πάρει το λόγο για κάποια πιο τεχνικά ερωτήματα. Λοιπόν, ε, προνομιακές σχέσεις με κάποια κράτη. Μίλησα όντω για τη, για Γαλλική Δημοκρατία και την Ιταλική Δημοκρατία που είναι οι δύο μεγάλες ε, γειτονικέ μας χώρες. Ε, είναι αμοιβώς επικερδής η εταιρική σχέση που έχει συγκροτηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες με αυτά τα δύο κράτη. Υπάρχουν πάρα πολλοί που διασχίζουν τα σύνορα και έρχονται καθημερινά στο πριγκιπάτο για να εργαστούν είμαστε, αν θέλετε, μια, μια δυναμική πηγή θέσεων εργασίας ε, για αυτούς τους ανθρώπους που ενδεχομένω ε, δεν θα έπαιρναν στην αγορά εργασίας στις ε, χώρες προέλευσής τους. Στις αγωγικές μου παρατηρήσεις σας μίλησα επίσης για το ε, ΦΠΑ και για το φόρο επί των κερδών, για το, σύστη, το γαλλικό σύστημα, δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση μονομερός να αυξομοιώσουμε τους συντελεστές, δεσμευόμεστα να εφαρμόσουμε τους εφαρμοστές γαλλικούς συντελεστές, όπως σας είπα εξάλλου συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ευρωστία και ε, στα ε, κέρδη και έσοδα του πριγκιπάτου. Διακόπτει ο Πρόεδρος, ε, επ' αυτού θα μου επιτρέψετε. λέτε ότι εφαρμόζεται γαλλικούς συντελεστές κατά τη διαστολή με άλλες, για, με άλλες χώρες. Δεν μπορείτε λοιπόν να τροποποιήσετε ε, για αυτούς τους δύο φόρους, τους συντελεστές. Όλοι ωραία. Λοιπόν, για τις φορολογικές συμφωνίες, γιατί αναφέρθηκε ο κύριος Έγγελ σε αυτό το ζήτημα και το συζητήσαμε και για άλλες φορολογικές αρχές, πάλι ακολουθείτε τη Γαλλία. Ε, μιλώ υπό τον έλεγχο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ε, φορολογικών υπηρεσιών ε, που θα δώσει πιο συγκεκριμένη απάντηση δεν κωδικοποιήσαμε βάσει του L81α και β την διαδικασία σύναψης φορολογικών συμφωνιών. Παρότι δεν ε, εξέλιψε αυτή η κωδικοποίηση, εφαρμόζουμε τις ε, ίδιες, του ίδιου τύπου ε, συμφωνίες και σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε έλλειψη απάντησης συστηματικά ε, λάβαμε ε, ε, τις ερωτήσεις και στείλαμε γραπτές απαντήσεις για την εφαρμογή αυτών των φορολογικών συμφωνιών. Υπουργός, ε, θα ήθελα να σχολιάσω κάτι σε με τα ιδρύματα, foundations, διότι αυτή την ερώτηση μας την υποβάλλουν συχνά. Έχουμε λιγοστά τέτοια ιδρύματα και ε, περίπου 20 και ο στόχος είναι κοινοφελής, είναι φιλανθρωπικοί οργανισμοί. Μπορώ να σας δώσω και τα ε, συγκεκριμένα στιγμή. 11 για ε, τη φιλανθρωπικού χαρακτήρα, 3 για τις υποτροφίες των φοιτητών, 3 για την επαγγελματική κατάρτιση και τα καλλιτεχνικά, την καλλιτεχνική δραστηριότητα, για τον αθλητισμό, για τα ζώα, αυτά ελέγχονται κάθε χρόνο και ο Υπουργό Οικονομικών ε, λαμβάνει ετησίω μία έκθεση για τη δραστηριότητά τους και μία ειδική επιτροπή όπου προεδρεύει ο ομόλογο μου για τις εσωτερικέ υποθέσεις ε, αλλά και ο υπεύθυνο για τι δικαστικές υπηρεσίες, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ελέγχουν ε, στη συνέχεια αυτέ τι εκθέσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως όταν συζητούμε για ιδρύματα σε εμά ε, διαφέρει κατά πολύ η κατάσταση διότι είναι ως επιτοπλίστων φιλανθρωπικοί οργανισμοί. Ε, το πλέον σημαντικό ενδεχομένως από αυτά που ακούσαμε είναι η προσέγγιση που ακολουθούμε για το BEPS και η υποστήριξη που προσφέρει σε αυτή την ε, πρωτοβουλία, σε αυτό το κίνημα, το Μονακό. Μην ξεχνάτε το μέγεθος τη διοίκησή μα και τον αριθμό των μεγάλων προτεραιοτήτων και προκλήσεων που αντιμετωπίσαμε. Ίσως δεν ήμασταν τόσο προδραστικοί, αν θέλετε, σε σχέση με άλλε χώρες, όμως ε, όταν ήρθε ο κύριος Μοσκοβισή στο Μονάκο επαναλάβαμε ότι υποστηρίζουμε ε, την πρωτοβουλία και της διατάξεις και εξάλλου τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, όπως είπανε και άλλοι συμμετέχοντες σε τις σημερινές ακρόασεις, θα έχετε καταλάβει πώς κάποιες επιπτώσεις σχετίζονται λιγότερο με το βιομηχανικό και κοινωνικό και τερικό ιστό ε, του πριγκιπάτου και γι' αυτό θα δείξαμε σε προτεραιότητα την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του πρωτοκόλλου που ε, επισυνάψαμε συμφωνία τον περασμένο μήνα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλειφθεί αυτό ως έλλειψη υποστήριξης από πλευράς μας. Μόνο ε, απαιτούμενη ιεράρχηση προτεραιοτήτων ε, των δράσεων που θα πρέπει να φέρουμε εις πέρας. Καλώς, σας ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο. Ο Φρανκ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, αλλά κύριε Υπουργέ, να επανέλθω σε κάτι. Θέλω να σας πω λοιπόν. Κάποιοι θα θυμούνται τα προβλήματα που είχατε με τη Γαλλία την αρχή της δεκαετίας του 60 και πώς οδηγηθήκατε στη διευθέτηση την τελωνιακή με τη Γαλλία τότε. Στην πράξη. Μια Ιταλική, μια Γαλλική επιχείρηση. Γιατί θα ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μονακό σαν οικονομικό χρηματιστικό κέντρο. Γιατί να δημιουργηθεί μια ανώνυμη εταιρεία στο Μονακό γιατί να έχει μια επιχείρηση παρουσία στο Μονακό. Αν δεν ε, οφείλεται αυτό το κίνητρο μόνο και μόνο σε φορολογικά κίνητρα. Αυτό που είπατε, ήδη δώσατε απάντηση στο τέλος ερωτήσεως, δεν έχει καμία σχέση με το φορολογικό ζήτημα. Φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι μόνιμοι κάτοικοι που διαμένουν στο Πριγκιπάτο, που ζουν στο Πριγκιπάτο, πολλοί είναι υπήκοοι χωρών της Ενώσεως και μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να θέλουν να δημιουργήσουν μια οντότητα στο Πριγκιπάτο του Μονακό που θα δραστηριοποιείται ίσως και εκτός του Πριγκιπάτου αλλά δεν επιλέγουν τον πριγκιπάτο για φορολογικούς λόγους. Η δραστηριότητα της επιχειρήσεως, οι περισσότερες είναι μικροεπιχειρήσεις. Είναι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στο Μονακό. Μεγάλη πλειοψηφία αυτών είναι φυσικά πρόσωπα, είναι οικογένειες, είναι άνθρωποι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις ε, ικανότητες τους, ε, τις δεξιότητες, τις γνώσεις τους που ανέπτυξαν κατά την καριέρα τους, να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες τους για δικό τους λογαριασμό ή να δημιουργήσουν μια επιχείρηση στον τομέα των υπηρεσιών, το βιομηχανικό τομέα, τον εμπορικό τομέα, για να παράξουν δραστηριότητα εκεί που βρίσκονται, εκεί που διαμένουν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης στις κοινότητες και τις περιοχές που γειτονεύουν. Αυτό είναι το κίνητρο παρά ε, το ότι διαλέγουν αυτή τη δικαιοδοσία για λόγους φορολογικούς. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο λόγος όπου ένας Ιταλός που δεν διαμένει στο Μονακό ή Γάλλος που ε, ε, δουλεύει στο Μονακό, το διαλέγει το Μονακό να εγκατασταθεί στο Μονακό για να θέλει για άλλους λόγους πέρα από την οποία να θέλει να αναπτύξει κάποια δραστηριότητα. Θα έλεγα, λέει ο Πρόεδρος, θα μιλήσουμε για τις πολυεθνικές το απόγευμα. Ακούσαμε 15 πέρσι και καμία της τις δεν έχει παρουσία στο Μονακό. Δυστυχώς για το Μονακό και για την ε, Ευρώπη. Καλώς, σας ευχαριστώ. Πάμε σε δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ο Μάρκο Βάλι για το EFTT έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ τα μέλη, τους εκπροσώπους των χωρών μάλλον αυτών που ήθελαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, οι απαντήσεις είναι πιο εξαντλητικές από άλλες. Απευθύνομαι προς τον εκπρόσωπο του Λίχτενστάιν γιατί μου διηγήθηκαν κάποιες αμφιβολίες. Είπε ότι υπάρχει δυνατότητα ε, να ε, δοθούν πληροφορίες από τις αρχές για τα καταπιστεύματα κλπ. Αν μια αρχή χρειάζεται τις πληροφορίες, πρέπει να υποβάλει αίτηση για να δοθούν οι πληροφορίες. Σε επίπεδο πολιτικό, Συζητείτε μια δυνατότητα να συλλεχθούν αυτές οι πληροφορίες και να υπάρχει επαφή με τις αρχές των άλλων χωρών για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ή παρέχονται οι πληροφορίες μόνο κατόπιν ετήματος για το θέμα των τραπεζών. Είναι σημαντικότατο θέμα. Πρόσφατα υπήρξε μια υπόθεση στην Ιταλία. Υπήρξε μια μεγάλη φοροδιαφυγή, τεράστια φοροδιαφυγή μεταξύ, το, από την κρατή Σουής που πουλήγε, πουλάγε ασφαλιστήρια συμβόλαια στο Λίχτεστάν. Το σκάνδαλο αφορούσε 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε φοροδιαφυγή. Ήτανε ψευτοσυμβόλαια ασφαλιστικά που έγιναν ε, μέσω Λίχτενστάιν. Γίνονται έρευνες. Προβλήθηκε πολύ στα μέσα ενημέρωση αυτή η υπόθεση. Σαν Λίχτενστάιν έχετε πρόθεση να λάβετε μέτρα στεφόμενη κατά ποιες ε, της τράπεζας αυτής που δημιούργησε κακή εικόνα για την χώρα. Υπάρχουν αυτές οι τράπεζες λοιπόν που ακολουθούν πρακτικές που δεν είναι καθόλου ηθικές. Εάν δεν στραφούμε εναντίον τους δεν θα καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να βασιστούμε σε αυτό το στόχο, να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο. Αλλιώς δεν θα νικήσουμε ποτέ τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή γιατί περνάνε αυτές οι ροές μέσω του τραπεζικού συστήματος. Μία ερώτηση που σχετίζεται με τον έλεγχο των τραπεζών. Η Ανδόρα και το Μοναχό υιοθετούν το ευρώ, αλλά είναι εκτός της εποπτείας, της ενιαίας εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γίνονται συζητήσεις, ούτω ώστε να υπάρχει εποπτεία αποτελεσματική, διότι έχουν τράπεζες που κάνουν μεγάλες επενδύσεις και μπορούν να είναι τράπεζες που είναι συστημικές. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Η Μπάρμπαρα Κάπελ έχει το λόγο. με τις ομάδες. Ευχαριστώ. Ε, Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους υψηλούς ε, εκπροσώπους των τριών πριγκιπάτων. 28 Ιανουαρίου εξέδωσε μια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας ενημερώνει για την εξωτερική στρατηγική για μια αποτελεσματική φορολόγηση που θα βασίζεται κυρίως σε συνέπεια και διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια για υπεύθυνη ε, δράση φορολογικά. Και αυτή η στρατηγική αφορά και τρίτες χώρες παρούσε σήμερα. Βέβαια στα φορολογικά ε, συστήματα υπάρχουν άλλα κριτήρια, διαφάνεια, ανταλλαγή πληροφοριών ε, και θεμητός φορολογικός ανταγωνισμός. Για τη διαφάνεια ακούστηκε και σήμερα, κατά κύριο λόγο μας ενδιαφέρει αυτόματη η ανταλλαγή απόψεων, δηλαδή ε, πληροφοριών μάλλον. Οι προδιαγραφές του ΩΣΑ να υιοθετηθούν αυτόματα. Εκατό κράτη ήδη έχουν δεσμευτεί και μεταξύ αυτών τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτόματα και επίσης ενημερώνουν για ε, φορολογικές συμφωνίες ε, διεθνούς ε, βεληνικούς για τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα από το 2017. Από εκεί και πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ακούστηκε υπάρχει υποχρεωτική αναφορά αναχώρα για τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα και ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο πρώτων υλών και στην δασοκομεία. Είπατε για την αυτόματη ανταλλαγή απόψε ε, ότι συγγνώμη πληροφοριών θα την ε, υιοθετήσετε και δεσμευτήκατε και οι τρει. Και θέλω να ρωτήσω κάτι την εκπρόσωπο του Λίχτενστάιν για τι εκθέσει αναχώρα. Έχετε επιφυλάξει για το δημόσιο χαρακτήρα. Αν κατάλαβα καλά από την εκπρόσωπο τη Ανδόρα, αυτό το καιρό ε, κάνετε μια εκτίμηση αντικτύπου, μελέτη επιπτώσεων δηλαδή. Στι εκθέσει αναχώρα, λοιπόν, ποια είναι η θέση του Μονακό, που δεν την άκουσα. Και δεύτερον, ποια είναι η θέση σα, του Μονακό πάντα, για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές συμφωνίες ε, και προκαταρκτικές συμφωνίες. Και δεύτερο, για το θεμητό φορολογικό ανταγωνισμό, το G20, ο, ο ΣΑ και οι παρούσες εδώ τρίτες χώρες έχουν συμφωνήσει να προσχωρήσουν στον ΠΕΠΣ για την καταπολέμηση της φορολογικής διάβρωσης, της διάβρωσης της βάσης και της ε, μετατόπισης των κερδών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι οθητήρια δύναμη εδώ, κινητήρια δύναμη, το δήλωσε πρόσφατο ο Επίτροπος Μοσκοβισή και πέρα από τα ΠΕΠΣ υπάρχει και κοινοτικό πακέτο μέτρων για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Πάντα φέτος το Γενάρη θα ε, κατάθεσε αυτά και ο κώδικας δεοντολογίας ενημερώνεται επίσης. Έρχομαι τώρα στην ερώτησή μου προς τους εκπροσώπου. Πρώτον, στον εκπρόσωπο του Μονακό, γιατί δεν κατάλαβα ακόμα από αυτά που είπατε πώς προτίθεστε ε, να εφαρμοστεί και πώς εφαρμόζεται αυτό τον καιρό το BEPS του ΟΣΑ, οι δύο εκπρόσωποι Ανδόρα και Λίχτενστάιν το είπαν πάρα πολύ συγκεκριμένα και μια ερώτηση και προ του τρει. Ε, το πακέτο μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πώς το βλέπετε το Ιανουαρίου του 2016 για παράδειγμα να ε, υπάρχει exit tax, switch over, να εκπίπτουν τα, οι φόροι και πάει λέγοντας το CFC και η εξουδετερώση ε, ε, υβριδικών ε, αναντιστοιχείων. Ευχαριστώ. Ο Παύλο Σάλβα ε, από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια πολύ απλή ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω τι ποσοστό των φορολογικών εσόδων της Ανδόρας Λίχτενστάιν και Μονακό προέρχονται από υπηρεσίες και προϊόντα που παράγονται στην επικράτειά σας. Και ποιο είναι το ποσοστό του φόρου επιχειρήσεων που προέρχονται από δραστηριότητες ε, εξωχώρης. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Απλή ερώτηση. Θέλω απαντήσεις. Λοιπόν, οι τους σοσιαλιστές Μανουέλ Μορέλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα απευθυνθώ προς την εκπρόσωπο του Λίχτενστάιν. Σε αυτά που είπε μας έλεγε ότι δεν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγματι. Είσαστε μέλος όμως του ΕΟΧ και της ΕΖΕΣ και του ΣΕΝΚΕΝ νομίζω αν θυμάμαι σωστά. Λοιπόν, εκεί είναι χώροι που εφαρμόζονται οι αρχές δημοκρατικές και της ισότητας. Ακούγοντάς σας, μου δημιουργήθηκε με ανησυχία. Φαίνεται να δέχεστε ότι ειδικεύεστε χαμηλή φορολόγηση και ότι δεν είναι πρόβλημα. Και δεχόσαστε το χαρακτηρισμό του φορολογικού παραδείσου στο διεθνές πλαίσιο. Διότι όμως αυτό οδηγεί σε φορολογικό ντόμπινγκ που καταπολεμούμε. Έχουμε με τρεις ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στα tax rulings. Τάξη μεγέθους. Πώς τέτοιες συμφωνίες γίνονται στο Λίχτενστάιν κάθε χρόνο, tax rulings. Αναφερθήκατε σταδιακή μεταρρύθμιση του EP Box. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα. Και επαναλαμβάνω και το ερώτημα του προλαλήσατε συναδέλφου. Πολύ ενδιαφέρον. Όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα, πόσα έσοδα αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που παράγονται, παρέχονται στο Λίχτενστάιν. Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε για την ίδια μάδα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα εγώ να απευθυνθώ στην Υφυπουργό Οικονομικών της Ανδόρας και να κάνω εξής τρία ερωτήματα. Πρώτον, εάν ισχύει ότι η φορολόγηση των επιχειρήσεων, ο συντελεστής δηλαδή είναι 10% με ελαφρύσεις και μειώσεις, κατά μέσο όρο για τις επιχειρήσεις ποιος είναι ο συντελεστής. Αν ισχύει ότι μη κάτοικοι δεν πληρώνουν για τα μερίσματα φόρο, δηλαδή μπορεί να έχουν λογαριασμούς χωρίς να φορολογούνται οι καταθέσεις τους, τραπεζικούς. Και αν ο φορολογικός συντελεστής royalties είναι 5%. Εάν ισχύει αυτή η πληροφορία, πρώτη ερώτηση, πιστεύετε ότι αυτό είναι τμήμα, πώς να το πω τώρα, μιας ε, φορολογικής πολιτικής ε, θεμητής και πιστής ε, με τις γειτονικέ σας χώρες. Ή μήπως αυτοί οι φορολογικοί συντελεστές ευνοούν την εγκατάσταση με τρόπο ε, τεχνητό ε, στην Ανδόρα Ισπανικών, για παράδειγμα, εταιριών. Εν τυχαίο παράδειγμα δανείζομαι. Δεύτερη ερώτηση. Μία από τις βασικές τράπεζες, η ιδιωτική τράπεζα Banco Privado de Andorra, κατηγορήθηκε ότι ξεπλένει χρήμα από παράνομε προστιδιότητες, από χώρε όπως είναι η Ρωσία και η Βενεζουέλα ιδιαίτερα. Το 2014 συνέβησαν όλα αυτά. Και ρωτώ, έχει ανδώρα φορολογική αστυνομία, η ε, ε, ΣΔΟΕ ας πούμε ή μια εποπτική αρχή για να εξασφαλίσει ότι τέτοια πράγματα δεν πρόκειται να επαναληφθούν. Γιατί εγώ αναγνωρίζω ότι είναι σε καλό δρόμο η ανδώρα και εκτιμώ και τις πολιτικές προθέσεις σας, κυρία Υφυπουργέ, αλλά ουσιαστικά αυτό που συνέβη με την τράπεζα αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και ερώτηση τρίτη τώρα. Στην Ισπανία δυστυχώ, μεταξύ των διαφόρων προβλημάτων που είχαμε διαφθορά, υπάρχει και ένα το οποίο ξεχωρίζει διότι η οικογένεια του Προέδρου ε, της Καταλωνίας του Περιφερειάρχη, του κυρίου Πουζόλ τότε, είχε στην Ανδόρα επί χρόνια πολλά ε, την περιουσία της. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ήταν, ε, πολλά τα λεφτά. Και μάθαμε, πρώτον από ό,τι φαίνεται γιατί ο ίδιο ο κύριος Πουζόλ όταν έκανε φορολογική αμνηστία το 2013 η Ισπανία αναγκάστηκε να αναγνωρίσει ότι είχε αυτά τα λεφτά στην Ανδόρα αλλά η δικαστική έρευνα μετά έδειξε η ανάκριση ότι δεκαετίες ολόκληρες είχαν λεφτά εκεί στην Ανδώρα. Μα ήταν περιφερειάρχης ο άνθρωπος, τόσο σημαντικής περιφέρειας όπως είναι η Καταλωνία. Και σας ρωτάω, ε, αυτό συνιστά φορολογική τώρα πίστη και αφοσίωση. Γιατί οι αρχές της Ανδόρας δεν ενημέρωσαν για την περιουσία που έκρυβε η ε, οικογένεια που Πουζόλ στην Ανδόρα. Γιατί δεν ενημερώσατε την Ισπανία. γιατί έχει θορυβηθεί ο κόσμος πάρα πολύ για την αξιοπιστία, ε, για το πόσο ε, είναι φορολογικά πιστή η Ανδόρα. Ξέρω ότι είστε σε καλό δρόμο, επαναλαμβάνω, και ξέρω ότι δημιουργήσατε τώρα μια εφορία. Εντάξει, πρόσφατα, όπως είπατε, ε, δημιουργήθηκε αυτή η φορολογική αρχή, αλλά είναι εκ των όνων κάνευ να καταλάβετε ότι πρέπει να διανύσετε αυτό το δρόμο γρήγορα. Και έτσι θα καταλάβετε και τις δικές μας αμφιβολίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Δεν μπήκε στο πεδίο των ερευνών μας αυτή η τελευταία σας παρατήρηση. Πολιτική φύση πολιτικής φύσης παρατήρηση, πολύ σημαντική, όμως ε, δεν σχετίζεται με αυτά που εξετάζουμε. Γόναν Λέρνερ από το ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε. 47.000 είναι περίπου οι επιχειρήσεις ε, στο Λίχτενστάιν. Αν ε, υπολόγισα σωστά, κάθε πολίτης λοιπόν έχει 1,27 εταιρείες ε, στο Λίχτενστάιν. Φυσικά πολλές είναι holding companies από μεγάλες πολυεθνικές ή από εταιρείες shell, δηλαδή μονομένων ιδιωτών. Ε, και ε, ε, πολλές χρησιμοποιούνται για φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή. Αλλιώς για ποιο λόγο να έχετε τόσες πολλές επιχειρήσεις στο Λίχτενστάιν. Εγώ δεν βρίσκω καμία άλλη λογική εξήγηση. Ας είμαστε λοιπόν ειλικρινείς. Χώρες όπως το Λίχτενστάιν φοηθούν τις πολυεθνικές στην φοροαποφυγή. Με ποιο τρόπο θέλετε να ενισχύσετε τη διαφάνεια του Δημοσίου Μητρώου όπου υπάρχουν πολλές ε, θηγατρικές ε, ε, μεγάλων πολυεθνικών όπως η ΚΕΑ παραδείγματος χάρη. Και το ίδιο ρωτώ και την Ανδόρα και το Μονακό. Έχετε φήμη ε, έλλειψης διαφάνειας στα δημόσια μητρώα επιχειρήσεων. Θα ήθελα να ξέρω πώς και πότε σκοπεύετε να ε, δώσετε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Φερέιρα, η Ελίζα από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Θέλω ε, να επανέλθω σε κάποια από τα ερωτήματα που έθεσαν ε, συνάδελφοι για την προνομιακή μεταχείριση του τραπεζικού τομέα από όλες τις χώρες που εκπροσωπούνται εδώ και όλος ιδιαίτερο από το Μονακό. Έχω μία πληροφορία, όχι κάποια μυστική πληροφορία, αλλά ενημερώθηκα ότι για τις γαλλικές ε, τράπεζες, παραδείγματο. χάρη, έχετε την BNP Paribas στο Μονακό με τζίρο 62 εκατομμύρια βάσει των λογαριασμών προφόρων και 22 εκατομμύρια αλλά δεν έχει καταβληθεί φόρος στο Μονακό για αυτά. Το ίδιο και είναι δημόσιες προφορίες αυτές για τις θηγατρικές της Société Γενεγάλ. Μπορείτε ξεκάθαρα να μας πείτε στον τροπεζικό τομέα ποια η σχέση σας με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης με ποια ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία έχετε συμμορφωθεί και με ποια όχι. Ξεκάθαρα πώς τοποθετήσετε σε σχέση με την κείμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία γιατί τώρα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ε, ε, στην, ε, στις εκθέσεις αναχώρα και στη διαφάνεια βάση του CRD και τη συνεργασία ανάμεσα στις τραπεζικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, ποια, ε, πώς συμπεριφέρεστε εν γέννη σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό τομέα και το τραπεζικό τομέα. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Ακούσαμε και πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις τώρα προς συγκεκριμένους συμμετοχούς. Κυρία Ντουρανή. Ευχαριστώ. try to, to make Θα προσπαθήσω να δώσω μια συνολική απάντηση. Πρώτα απ' όλα για τη νομισματική συμφωνία και τον, ε, την εποπτεία των τραπεζών. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας Έχουμε σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Περιπίν, πρέπει να δίνουμε στατιστικά δεδομένα και υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών με την ΕΚΤ. Είναι σημαντικό αυτό, διότι δίνουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Όπως ξέρετε, σε όλες τις οδηγίες πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το μέγεθος κάθε χώρας. Άλλο να είναι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και άλλο μικρότερες επιχειρήσεις. Αυτό κάνουμε τώρα. Συζητούμε και με την έκτη για να δούμε αν με αυτές τις πληροφορίες θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία για, το, ε, για την κάθε χώρα. Για την εποπτεία έχουμε έναν επόπτη με εποπτική αρχή και Δεν μας υποπτεύει εμά κανείς, αλλά μας είπαν ότι αν ε, χρειάζεται συντονισμός ε, υπάρχει ανοιχτή γραμμή με το, την ΕΚΤ. Δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα με στην επαφή με την ΕΚΤ. Ζητούμε εμείς περισσότερα, περισσότερη πρόσβαση πληροφορίες ε, της ΕΚΤ. Φυσικά όταν κάποιος έχει αυξημένες υποχρεώσεις θέλει και αυξημένα δικαιώματα. Ε, για να έχει περισσότερες πληροφορίες. Προβλέπονται όμως όλα αυτά και ήδη συζητούμε σε μια μεικτή επιτροπή που έχουμε με τους εκπροσώπους όλων αυτών των θεσμικών οργάνων. Με την έκτη είμαστε σε άμεση επαφή και αν χρειαστούν επισκέψεις επί τόπου τις κάνουμε και αυτές Κάνα πρόβλημα. Σε σχέση με το δημοσιοοικονομικό και φορολογικό πλαίσιο. Δεν εφήβραμε τίποτα εμείς. Βλέπαμε τι ίσχυε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο. Ποιο είναι... Είναι καλό το σύστημά μας. Ο στόχος δεν είναι φορά Το πλαίσιο, το πλαίσιο αυτό, όπως έλεγα, μας επιτρέπει να φτιάξουμε τη νέα ανδώρα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε 8 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο για τις ε, εταιρείε πληροφορικής. Για τον ε, τομέα της υγείας, ε, γιατί είμαστε και στα βουνά, για την παιδεία. Εμείς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό των επισκεπτών, των τουριστών. Γι' αυτό έρχονται οι επιχειρήσεις στην Ανδώρα και όχι για την ε, φοροαποφυγή, γιατί έχουν αυτές τις νέες δυνατότητες. Θυμηθείτε επίσης ότι είναι μικρές επιχειρήσεις αυτές που έρχονται. Μεγάλες δεν έχουμε. Πέντε άτομα προσωπικό είναι μικρομεσαίες. Παρόλα αυτά εμείς παρακολουθούμε τον ΠΕΠΣ και τις εξελίξεις κατόπιν αιτήματο ανταλλαγή, αυτόματη ανταλλαγή προφορών εξελίξεις υπάρχουν. Το σημαντικό είναι να γίνει το πρώτο βήμα. Και εγώ πιστεύω ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Ε, θα χρειαστούν ίσως προσαρμογές. Κάθε φορά πάντως λαμβάνουμε αποφάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, προς συμφέρον της χώρας, όχι για να ενισχύσουμε τη φορά αποφυγή. Για να ενισχύσουμε το ειδικό βάρος σαν δώρο σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Για τα CDAs, για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, δεν είχε κανένας από τους εταίρους μας πρόβλημα και για ε, τη ρήτρα κατά των καταχρήσεων και αυτά. Δεν, ε, τα, τα υπογράψαμε τις συμφωνίες. Κοιτάξτε, τα τελευταία δύο χρόνια υπογράψαμε όλες τις ιδιές μας. Τα λέω αυτά για να ε, τεκμηριώσω το ότι δεν ε, είναι ε, προβληματικό το φορολογικό μας σύστημα και όλα τα κάνουμε στην εργασία με άλλες χώρες. Τώρα, με ρωτήσατε για το 10% εταιρικό φόρος για τα ρόγελ της, για τους μη διαμένοντες δεν το καθεξής. Ο ονομαστικός ε, συντελεστής σχεδόν ταυτίζεται με τον πραγματικό. 9 έως 10%. Αυτός είναι ο φυσιολογικός ο συνθέστερος συντελεστής για τους μη διαμένους μπορεί να υπάρξει διαφορά αλλά και για τα μερίσματα πρέπει να είναι ε, δική μας επιχείρηση και δεν ισχύει για όλους, για τα ρόγιαλ της μπορεί να υπάρξουν κάποια προνόμια, όμως συγκρίσιμα με αυτά που βλέπουμε σε άλλες επιχειρήσεις, τίποτα εξαιρετικό. Και ξαναλέω, το ότι έρχονται οι επιχειρήσεις δεν οφείλεται σε αυτό, αλλά στις ιδιαιτερότητες της χώρας μας, διότι ε, έχετε το τραπεζικό τομέα, τους τουρίστες, ε, τα 8 εκατομμύρια που σας έλεγα τουρίστες το χρόνο, Αυτά ψάχνουν οι επιχειρήσεις ε, γιατί στον τομέα της υγείας παραδείγματος χάρη θέλετε να κάνετε μία εγχείρηση και ε, οι συγγενείς πάνε για σκι ενώ εσείς είστε στο νοσοκομείο. Για το τραπεζικό τομέα. Σας είπα ότι έχουμε το WIFAN, τον επόπτη για το, την νομοποίηση ε, των παρανόμων εσόδων και τον... Ε, τον οικονομικό επόπτη. Δεν είναι και τίποτα καινούριο αυτό. Υπάρχει και, και παρακολουθούμε όπως και άλλες οι χώρες τις αξιολογήσεις ε, για το, την νομοποίηση εσόδων. Είμαστε στο πέμπτο γύρο αξιολογήσεων. Συμμετέχουμε και στον Ιόσκο. Μας, ε, μας παρακολουθούν. Αν δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις δεν είσαστε μέλος Συμφωνίων Ιόσκο. Στην Νομισματική Συμφωνία στο παράρτημα έχετε σειρά οδηγιών με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθείτε. Πριν από τον BPA. τα είχαμε εμεί όλα αυτά στην νομοθεσία μας. Κανένα πρόβλημα δεν είχαμε. Και για την ή για αυτή την τράπεζα, υπήρχε θέμα με τη διοίκηση, όχι με την ίδια την τράπεζα. Συμβαίνουν αυτά. Όχι ότι είναι φυσιολογικά, αλλά συμβαίνουν και στις καλύτερες χώρες. Δεν μπορούμε να τους ελέγχουμε όλους όλη την ώρα. Μπορούμε να το δούμε και θετικά πέρσι. Όλα τα βήματα έγιναν. Το Φεβρουάριο με την αξιολόγηση αναφέραν αυτό ότι η κυβέρνησή μας έχει κάνει ε, όλες τις απαιτούμενες Όχι Όχι δεν έχουμε εποπτικές αρχές, το αντίθετο έχουμε και είναι πάρα πολύ καλή δουλειά που κάνουν. Και σε σχέση με αυτό που δημοσιεύτηκε στη ΣΥΠΑ τα λέω αυτά. Ξέρετε, για μας είναι απαραίτητο για να ε, έχουμε μεγαλύτερη εξοπιστία για την κυβέρνηση και για τις εποπτικές αρχές, ε, για τις, ε, τα rating agencies, επιχειρήσεις αξιολόγησης, το, το αναφέρουν αυτό. Για τα δικαστικά ε, ζητήματα, ε, να σας πω ότι όταν υπήρξε δικαστική απόφαση, τις δώσαμε τις πληροφορίες, αλλά τέτοια υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Δεν, δεν είναι δική μας αποκλειστικότητα. Και τώρα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και γίνεται αυτό που πρέπει. Δεν έχω προσθέσω τίποτα. Παρακολουθούμε τα βήματα που κάνουμε. Και μην ξεχνάτε ότι σε αυτό το σημείωμα λένε οι ΙΠΑ ότι κάνουμε τις προσπάθειες που πρέπει. Έχουν, έχουμε εξηγήσει όλη τη στρατηγική που ακολουθούμε. Και όπως σας είπα στην εισαγωγή μου, ό,τι χρειάζεται το κάνουμε. Δεν με τη... Βλέπουμε τις πρακτικές των υπολείπων ε, σε παγκόσμια κλίμακα μαθαίνουμε τα νέα από τον ΩΣΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλους τους διεθνείς οργανισμούς, αναλύουμε την κατάσταση και ευθυγραμμιζόμαστε αναλαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα. Πρόεδρος. Μπορείτε τώρα ή εν συνεχεία να απαντήσετε στην ερώτηση του Πάμπλο Σάλμπακ που αναφερόταν στα τρία πριγκιπάτα. Μπορείτε να μας δώσετε στοιχεία όσον αφορά το τζίρο που πραγματοποιείται στην Ανδόρα από επιχειρήσεις καταγωγής που προέρχονται την Ανδόρα και τον τζίρου των ε, ξένων επιχειρήσεων. Να συγκρίνουμε λοιπόν το δυναμικό που έχει κάθε δικαιοδοσία, κάθε κράτος και να δούμε πόσο ελκυστική είναι η κάθε χώρα. Αν δεν έχετε στοιχεία τώρα, μας τα στέλνετε γραπτός. Στρέφ, στρέφομαι προς το Λίχτενστάιν τώρα. Γκάι. Η ε, κυρία Γκάι έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σχετικά με το τελευταίο ερώτημα για τα στοιχεία. Δεν κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ εισοδήματο που παράγεται στο Λίχτενστάιν και εκτός Λίχτενστάιν. Άρα δεν μπορώ να σας δώσω στατιστικά στοιχεία αυτή τη στιγμή. Κάποιες ενδείξεις ίσως. Στην αρχική μου παρέμβαση αναφέρθηκα στη βιομηχανία, στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Οι πολύ μεγάλες βιομηχανικές μας επιχειρήσεις είναι οικογενειακές. ανήκουν σε κατοίκους του Λίχτενστάιν ή πολίτες του Λίχτενστάιν, φορολογούμενους, μεγάλους φορολογούμενους στο Λίχτενστάιν. Ένα παράδειγμα δίνω. Δεν μπορώ να σας δώσω όμως ιδιαίτερα συγκεκριμένα στοιχεία. Πιθανότατα, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, μπορώ από το εξή. να ξεκαθαρίσω ποιο είναι το καθεστώς της χώρας μου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτής. Παρέχονται οι πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Αυτά είναι τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Για συγκεκριμένη υπόθεση φοροδιαφυγής, απάτης κλπ που αφορά κάποια φορολογική αρχή κράτους μέλους, αν υποβληθεί αίτημα, το Liechtenstein συλλέγει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, πραγματικό ιδιοκτήτη εταιριών, ιδρυμάτων, καταπιστευμάτων, συλλέγουμε πληροφορίες για τα λογιστικά στοιχεία, για, τα, για τις τράπεζες, για τις συναλλαγές, Πληροφορίε που απαιτούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και στα πλαίσια των συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση του Global Forum, όπως σας είπα, ε, αναφέρονται στατιστικά στοιχεία για την ανταλλαγή πληροφοριών με τους εταίρους μας. Συμπελαμβανομένοι της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας, επί παραδείγματι. Μέχρι τώρα αυτή είναι η βασική μας εταίρη στην Ευρώπη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ένας από τους βασικούς μας εταίρους εκτός Ευρώπης. Πέραν αυτού, από το φορολογικό έτος 2016 θα αρχίσει η ανταλλαγή χρηματοπιστωτικών λογιστικών στοιχείων και όσον αφορά τις διαδικασίες συμμόρφωσης και διαδικασίες συλλογής πληροφοριών που αφορούν τα φορολογικά, όλα αυτά ξεκίνησαν σαν προσπάθειες τώρα. Όχι μόνο έχουμε λάβει δεσμεύσεις για την ορθή χρηστή επιμέλεια, ήδη εφαρμόζουμε λοιπόν τους σχετικούς κανονισμούς. Αντίθετα με άλλους παρόντες εδώ, εμείς κινηθήκαμε σε πολύ αρχικό στάδιο, από τους πρώτους. Δεν ανταλλάσσουμε μόνο πληροφορίες αυτομάτως, από το 2018 και πέρα, αλλά ήδη τώρα, μάλλον από του χρόνου, θα γίνει την αλλαγή πληροφοριών με όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι θα λαμβάνετε πληροφορίες για τα χρηματοπιστωτικά θέματα και για τους λογαριασμούς Ευρωπαίων που διαμένουν ε, στο Λίχτενστάιν και έχουν κάποια συμφέροντα σε κάποιο ίδρυμα στο Λίχτενστάιν. Η υπόθεση που αναφέρθηκε μιας ελβετικής τράπεζας αυτή είναι μια υπόθεση που τελεί έρευνα ακόμα. Δεν έχω λεπτομέρειες στη διάθεσή μου. Αν πράγματι ένα ασφαλιστικό προϊόν του Λίχτενστάιν χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς φόρο διαφυγής, αυτό είναι πολύ λυπηρό. Και το μόνο που μπορώ να πω σε αυτή τη φάση είναι να σας διαβεβαιώσω ότι αν μια τέτοια υπόθεση αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών από, που θα υποβληθεί στις Ιταλικές Αρχές, τότε βεβαίως το αίτημα αυτό θα αντιμετωπιστεί βάσει της συμφωνίας που δεσμεύει η Ιταλία και η Λίχτενστάιν. Μετά, Υπήρξε μια άλλη ερώτηση που ετέθη και αυτή αφορούσε τα μέτρα που προτάθηκαν να εφαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα BEPS του ΟΣΑ. Έχει δεσμευτεί το Λίχτενστάιν. Έχει συμφωνήσει να εφαρμόσει μια πρώτη δέσμη μέτρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΑ για τα ΜΠΕΠΣ. Θα κινηθούμε βάσει των προδιαγραφών ΟΣΑ και όχι βάσει του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι αυτό το κεκτημένο δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο Λίχτενστάιν βάση του παρόντος πλαισίου των συνθήκων. Αναφερθήκατε στην εξωτερική στρατηγική. Θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο. Τα εφαρμοστικά μέτρα και το σχέδιο οδηγίας που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου οδηγία σε σχέση με τις συστάσεις του ΩΣΑ εμείς καλωσορίζουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει επίσης τα BEPS Αυτό που θα αναμέναμε θα ήταν ότι τουλάχιστον εν μέρη σύμφωνα με το σχέδιο οδηγίας θα πρέπει η οδηγία να εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα δικαιώματα και υποχρεώσεις θα γίνονται σεβαστά στα πλαίσια της συμφωνίας ΕΟΧ. Και θα πρέπει να τα λάβει υπόψη και ο νομοθέτης Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δηλαδή, η θέση του Λίχτενστάιν σαν μέρος του ΕΟΧ όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων θα λαμβάνεται υπόψη. Αναφερθήκατε στο CFC ρήτρα εξόδου κλπ. Εμείς θα αναμέναμε αυτοί οι κανόνες να θεσπιστούν με βάση τη συμφωνία ΕΟΧ και με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συμφωνία μας. Η εξωτερική στρατηγική που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς θεσπίζει κριτήρια σαφή και αντικειμενικά. Το στηρίζουμε εν γέννη αυτό και ένθερμα. Σαφή αντικειμενικά κριτήρια. Και να υπάρξει και διάλογος με τις χώρες εταίρους. Το Λίχτενστάιν θεωρεί ότι είναι προνομιούχος εταίρος σαν μέλος του ΕΟΧ και εδώ και πολλά χρόνια έχει ξεκινήσει διάλογος όσον αφορά το θέμα του δεντρολογικού κώδικα για τη φορολόγηση επιχειρήσεων. Και θεωρούμε ότι θα συνεχιστεί αυτός ο διάλογος επί ουδετέρας βάσεως. Ετέθη άλλο ερώτημα. Αυτό αφορούσε τις φορολογικές συμφωνίες, τα tax rulings κατά πόσο το Λίχτενστάιν ακολουθεί αυτή την πρακτική και πόσες τέτοιες συμφωνίες συνάπτονται κάθε χρόνο. Προανέφερα ότι η φορολογική αρχή του Λίχτενστάιν εκδίδει αυτά τα rulings που ελέγχονται από την ΕΣΑ που είναι η υποπτική αρχή της ΕΖΕΣ κατά πόσο συμμορφώνονται με τη συμφωνία ΕΟΧ και κυρίως με τις διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων. Πόσα rulings εκδίδονται, περίπου 10 τέτοιες αποφάσεις το χρόνο, ισχύουν πενταετία κατ' εξαίρεση ίσως ισχύσουν, ίσως ισχύσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. τέτοιε αποφάσεις, τέτοια rulings μπορούν να εφαρμόζονται συνεχώ εάν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη στη φορολογική μας νομοθεσία. Καμία τέτοια απόφαση δεν μπορεί να εφαρμοστεί που αντιβαίνει τον νόμο. Και αυτό έχει εξακριβωθεί από το εποπτικό όργανο, την εποπτική αρχή. Η μεταρρύθμιση του IP, POX, του Patent POX, έχουμε αξιολογήσει τις συστάσεις του ΩΣΑ και τις σχετικές δράσεις στα πλαίσια αυτών των patent boxes εξακολουθεί το παρόν patent box που χρησιμοποιούμε να ισχύει μετά την μεταβατική περίοδο που θεωρείται αποδεκτή γι' αυτό σταδιακά θα εξαλειφθεί θα εξαλειφθούν αυτά τα patent boxes εκτός του προβλεπομένου χρονικού ορίου δηλαδή μέχρι το τέλος του 2020, κατά πόσο στο μέλλον ο η φορολογική νομοθεσία του Λίχτενστάιν θα προβλέπει την ύπαρξη ενός IP box που θα πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσει του ΟΣΑ, αυτό θα πρέπει να εξεταστεί. Θα αποφασιστεί. Μετά από αυτή την περίοδο θα δούμε κατά πόσο θα υπάρχει IP Box που συνάδει με το πλαίσιο του ΩΣΑ. Η άλλη επιλογή θα είναι να καταργηθεί αυτό. Uh, λοιπόν και κάτι άλλο όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων στο Λίχτενστάιν είναι ο ίδιος αριθμός που αντιστοιχεί στους πολίτες. Το Λίχτενστάιν δεν είναι ούτου ήταν ποτέ ένας επιχειρηματικός τόπος γνωστός χρησιμοποιούμενος για πολυεθνικές και δομές holdings. ούτε κατά παρελθόν. Ίσως μεταξύ άλλων διότι η φορολογική νομοθεσία του Λίχτενστάιν για τέτοιες δομές δεν ήταν ε, ελκυστική. Το ότι εταιρείες μπορούν να ιδρυθούν, να εγκατασταθούν σε κάποια άλλη ε, χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή χώρα ΕΟΧ, αυτή είναι η βάση της κοινή αγοράς. Άρα είναι κάτι που προωθούσε πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιθανότατα κατά το παρελθόν ίσως να υπήρξαν περιπτώσεις, κάποιες περιπτώσεις όπου τέτοιες εταιρείες εγκαταστάθηκαν και ιδρύθηκαν για να αποφύγουν φόρους ίσως να ισχύει κάτι τέτοιο αλλά μόνο κατά το παρελθόν δεν αφορά το παρόν κυρίως από όταν το Λίχτενστάιν δεσμεύτηκε το 2009 να ανταλλάσσει πληροφορίες κατόπιν ετήματος και το 2014 συμφώνησε για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και η δημιουργία εταιρεία ή άλλου νομικού προσώπου μόνο και μόνο για φόρο διαφυγή αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανέφικτο πια. Γιατί να συστήσει κανείς μια εταιρεία στο Λίχτενστάιν. Το Λίχτενστάιν είναι πολύ σταθερό είναι πολύ ελκυστικό σαν γεωγραφική θέση στην Ευρώπη. Standard και Poor's επιβεβαίωσε τη βαθμολόγησή μας του τριπλού αλφα. Δεν υπάρχει κρατικό χρέος. Υπάρχει πολύ υγιές σύστημα και πλαίσιο. Υπάρχει αξιόπιστο θεσμικό σύστημα, δικαιοσύνη, σωστή νομοθεσία ανήκουμε σε δύο οικονομικούς χώρους. Όχι μόνο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με την Ελβετία έχουμε το ελβετικό φράγκο σαν εθνικό νόμισμα και για καλό και για κακό δεν είναι και τόσο καλό τώρα η χρηματοστητική αγορά η αρμόδια αρχή της χρηματοστητικής αγοράς είναι ισχυρότατος φορέας συμμορφώνεται με ευρωπαϊκές προδιαγραφές Άρα το γενικό πλαίσιο για τη δημιουργία μιας επιχειρήσεως στο Λίχτενστάιν στην Ευρώπη είναι πολύ ελκυστικό. Η φορολογική νομοθεσία ίσως να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δημιουργείται μια εταιρεία στο Λίχτενστάιν. αλλά σήμερα δεν είναι ο μόνος λόγος λόγω της ανταλλαγής πληροφοριών. Άρα δεν είναι μόνο το φορολογικό καθεστώς αποκλειστικός λόγος δημιουργίας μιας επιχείρησης στο Λίθασταν πια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και στο Μονακό. Ε, δέχτη πάλι πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω και εγώ συγκεκριμένα όσο και σύντομα. Σε ό,τι αφορά το BEPS αναφέρθηκα προηγουμένως στο ζήτημα και στην ανακοίνωση του Επιτρόπου κυρίου Μοσκοβησής 28 Ιανουαρίου. Ε, ε, είπα ότι είχα την ευκαιρία να το συζητήσω μαζί τους 22 Φεβρουαρίου που ήρθε στο Μονακό και είναι μια πρωτοβουλία που εμείς υποστηρίζουμε και προσυπογράφουμε για τους λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως δεν ήμασταν τόσο πρόδραστοι εκεί σε αυτό το τομέα, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να σας ε, κάνει να πιστεύετε ότι αδιαφορούμε για το θέμα, το αντίθετο μάλιστα, ούτε ότι δεν έχουμε την πρόθεση να εμπλακούμε στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Όπως κάναμε και με πάρα πολλά σημεία που ακούσαμε για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών είτε στα πλαίσια του ΟΣΑ είτε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν υπάρχει ένα πεδίο με ίσους κανόνες παιχνιδιού και ακολουθούν όλες οι χώρες και το ε, πριγκιπάτο δεν μένει εκτός αυτής της προσπάθειας. Ε, αναφέρθηκε το MRU και MR, MSU. Ε, εμείς δεν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πήραμε επιστολή το 2015 που μας είπαν ότι ε, δεν μπορεί να βρει εφαρμογή σε εσά. Άρα δεν είναι ότι εμείς δεν το επιθυμούμε, αλλά σωστά προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε ότι δεν ισχύει για το Μονακό. Αλλά στη Συμφωνία Σύνδεσης που έχουν ε, αυτό το καιρό στη διαπραγμάτευση αρχές ε, του Μονακό ε, με την Κομισιόν και για το Άγιο Μαρίνο και την Ανδόρα ισχύει αυτό για την ενιαία εποπτική αρχή ε, στην Ευρωπαϊκή, αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τις τράπεζες που εδρεύουν στο Μονακό. Όταν όμως ε, μιλάμε για συστημικό κίνδυνο θα πρέπει να τονίσω ότι όλες οι τράπεζες που εδρεύουν σε εμά είναι υποκαταστήματα ή θηγατρικές μεγάλων διεθνών ομίλων. Ε, δεν υπάρχει ουσιαστικά τράπεζα του Μονακό που θα μπορούσε να σημάνει συστημικό κίνδυνο για το τραπεζικό μας και το οικονομικό μας σύστημα. Πολύτε περισσότερο, δεν υπάρχει συστημικός κίνδυνος για την Ευρώπη ή για το εξωτερικό του Μονακό. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι θυγατρικές μεγάλων ε, ομίλων ε, χρηματοπιστωτικών και ιδρυμάτων. Για τα φορολογικά έσοδα μπορώ να σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Για το ΦΥΠΙΑ που παράγεται ε, στο Μονακό και αφορά την κατανάλωση δηλαδή στο Πριγκιπάτο ή την ε, αγορά, αγοραπολισίες ε, διαμερισμάτων είναι 80% του συνόλου των φορολογικών εσόδων από το ΦΠΑ. Αντίστοιχα, ο φόρος επί των κερδών παράγεται από τις επιχειρήσεις που έχουν ε, τουλάχιστον 75% του κύκλου εργασιών στο πριγκιπάτο. Υπάρχει πραγματική οικονομική δραστηριότητα η οποία φορολογείται και χρησιμοποιείται ως βάση για να υπολογίζονται τα φορολογικά έσοδα και τα έσοδα του προϋπολογισμού του πριγκιπάτου. Ο αριθμός των επιχειρήσεων, σας τον ανέφερα, είναι κάποιες χιλιάδες, αλλά κυρίως πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, με ε, ε, ανθρώπους που ζουν, που διαμένουν μόνιμα στο Μονακό, έχουν μια δραστηριότητα και παράγουν κέρδη και για το κράτος. Έσοδα. Τονίζω ότι από το 1946 οι holding απαγορεύονται στο πριγκιπάτο του Μονακό. Ε, οι όμιλοι χαρτοφυλακίου, δηλαδή να μην εδρεύουν εταιρείε που να μην έχουν πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Αυτό απαγορεύεται στο Μονακό. Και δεν συμβαίνει. Ε, και το τελευταίο που με ρωτήσατε αφορά το φόρο των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα τη συνεισφορά κάποιων τραπεζών, ιδιαίτερα γαλλικών τραπεζών. Ε, τονίζω ότι μπορεί τα στοιχεία που να ακούστηκαν να μην ε, ήταν τελείως ενημερωμένα, διότι ο φόρος επί των κερδών είναι περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ στο Μονακό και οι τράπεζε είναι ο παριθμόν ένα συνεισφέρον για το φόρο των επιχειρήσεων. Μετά υπάρχουν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής και μία από τις τράπεζες που αναφέρθηκε πέρσι ήταν ο τέταρτος φορολογούμενος ε, που ε, καταβάλουν οι τράπεζες επί των κερδών τους. Δηλαδή σήμερα πραγματικά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ε, φόρου αυτού που πληρώνουν οι τράπεζες που, έχουν, ε, που είναι είτε φυγατρικές μεγάλων γαλλικών τραπεζών είτε άλλων ξένων τραπεζών. Αυτά είναι στοιχεία του 2015 που έχω στη διάθεσή μου. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ και εγώ. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Κατσδιάη, δεν ξέρω, εκτός καταλόγου ή κάποιοι συνάδελφοι που έκαναν ερωτήσει και θέλουν διευκρινήσεις συμπληρωματικέ επιπλέον θέματα. Ορίστε, ο Μπέρντ Λούκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι την εκπρόσωπο της Ανόρας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υφυπουργέ για την απάντησή σας προηγουμένως σε αυτό που σας ρώτησα. και αφορούσε τους φορολογικούς συντελεστές. Αλλά αυτό που είχα ρωτήσει εγώ κυρίως ήταν τι σας εμποδίζει εσάς στα πλαίσια αυτών των εξετάσεων στις οποίες προβαίνετε και στους ελέγχους τι βλέπετε να σας εμποδίζει να συνεργάζεστε στην τεκμηρίωση για τις τιμές μεταφοράς ε, ε, και μεταβιβάσεις. Και στην ε, έκθεση αναχώρα είπατε ότι το ελέγχετε, αν θα μπορέσετε να το εφαρμόσετε, αλλά δεν μπήκατε σε λεπτομέρειες. Ποια είναι τα υπέρ και ποια είναι τα κατά. Ωραία, το ελέγχετε. Έχετε εντοπίσει υπέρ και κατά μέχρι στιγμής. Και θα ήθελα να σας κάνω και άλλη ερώτηση. Στην, ε, εισαγωγή σας είπατε, συγγνώμη, ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί την Ανδόρα ως μη συνεργάσιμη ή ότι ε, έχει μικρή προθυμία. Τι σας ε, προσάπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς το δικαιολογεί αυτό, γιατί σας κατατάσσει έτσι. Ευχαριστώ, απάντηση. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο σημείο, ότι ε, μας κατατάσσουν στους μη συνεργάσιμους. Αυτό δεν είναι σωστό δίκαιο γιατί ακολουθούμε και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και όλες τις οδηγίες, ε, τις νομισματικές συμφωνίες ε, στα παραδείγματά μας. Επίσης έχουμε και μια νέα συμφωνία σύνθεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κάνουμε όλα αυτά διότι θέλουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε η χώρα να συμμορφωθεί όπως και οι υπόλοιπες. Είμαστε μικρή χώρα, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν θέλω να το επαναλάβω, αλλά θέλουμε να έχουμε μια ανοιχτή οικονομία, ένα νέο φορολογικό μοντέλο, να αλλάξουν ε, όλες αυτές οι καταστάσεις και να επέλθει διαφάνεια. Είναι πολλά αυτά που κάνουμε και δεν είναι καθόλου εύκολο. Είμαστε μικρή χώρα και λίγοι κάτοικοι. Ε, πηγαίνουμε σε όλες τις συνεδριάσεις, αναλύουμε τα πάντα. Δεν είναι δίκαιη αυτή η κατάταξη. Προσχωρούμε σε όλες τις συμφωνίες, συζητούμε τα πάντα. Γιατί μας προσάπτουν προθυμία. Σας είπα και προηγουμένως. Έχουμε το φορο, οι εταιρείε φορολογούνται εκεί που παράγουν το κέρδος. Δεν κάνουμε τίποτα περίεργο εμείς, τίποτα μυστήριο. Και οι συμφωνίες που έχουμε είναι διμερείς. Δεν τις υπογράφουμε μόνοι μας, υπάρχει και αντισυμβαλόμενο μέρος. Και είναι άδικο αυτό γιατί κάνουμε πολλές προσπάθειες. Τώρα, αυτό είναι δύσκολο για μας γιατί συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ΟΣΑ. Όταν πάω στο κοινοβούλιο μου και λέω όλα αυτά που κάνουμε, γιατί πηγαίνω στην Οικονομική Επιτροπή και εξηγώ τι κάνουμε και μετά βγαίνουν αυτές οι λίστες και σου λένε γιατί είσαι σε μαύρη λίστα αφού τα κάνεις όλα καλά, ε? κάτι τρέχει. Είναι σημαντικό για τη χώρα αυτό να αναγνωρίζεται και θα συνεχίσουμε να το λέμε πάντα. Σε ό,τι αφορά αυτά που κάνουμε ή που πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Ε, ξέρετε ότι κάνουμε τις διάφορες αξιολογήσεις, τις παρακολουθούμε, λαμβάνουμε υπόψη όλες τις συστάσεις που γίνονται και προσπαθούμε να βρούμε ένα καλό τρόπο να το κάνουμε. Τώρα είμαστε και στην ομάδα BEPS και αναλύουμε τι μπορεί να γίνει όταν συζητάτε για τις εταιρείες και τον εταιρικό φόρο. Πρέπει να πούμε και έχει σημασία αυτό το εξή. Οι εταιρείε που πληρώνουν φόρο είναι εταιρείε τη Ανδόρα. Αν είσαι ξένη εταιρεία και παρέχει υπηρεσίε στην Ανδόρα, ε, πληρώνει 10% που είναι ο φόρο για του μη κατοίκου. Έχουμε ειδικό καθεστώ για τον εταιρικό φόρο, ναι, έχουμε, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτό που αναλύουμε είναι αυτό πώς ε, επιδρά όλα τα υπόλοιπα, όλη την οικονομία αλλά και διεθνώς τι επιπτώσεις υπάρχουν. Δεν ξέρω αν θέλετε, έχω τα στοιχεία. Τι αντιπροσωπεύει ο φόρος ε, για τον προϋπολογισμό μας. Μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία για να έχετε μια καλύτερη εικόνα. Δεν ξέρω αν θα σας βοηθήσει. Με χαρά να το κάνω. Προσπαθώ να τα βρω κιόλα. Για να είναι πιο εύκολο να το διαπιστώσετε. Πρέπει να σας πω ότι για το 2015 είναι πρόβλεψη. Δεν είναι τα στοιχεία αυτά οριστικά. Για τους άμεσους φόρους πάνω κάτω έχουμε 69 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, από τις εταιρείε είναι τα μισά, 30. Και λάβετε υπόψη ότι μέσα σε αυτά και είναι και ο φόρος ε, από το τραπεζικό σύστημα που είναι 9%. Ε, επίσης, αν δείτε τώρα το φόρο εισοδήματος για τις οικονομικές δραστηριότητες, είναι η πρόβλεψη γύρω στα 20 εκατομμύρια. και για τη φορολόγηση των μη μόνιμων κατοίκων είναι 16. I mean, you can see more or less what is the, the percentage. Και τα υπόλοιπα είναι μάλλον αμεληταία. Λοιπόν, βλέπετε το ποσοστό αυτό. Και στις εταιρείε είναι 38 με τις τράπεζες μέσα. Στους έμεσους φόρους τώρα, ε, που είναι ΦΠΑ περίπου, 121 εκατομμύρια. Το διπλάσιο περίπου. Είμαστε μια χώρα που δεν εξάγουμε, αλλά εισάγουμε Είναι και αυτό μέσα. The taxes, that is one. Και έχουμε και άλλους φόρους που είναι 100 εκατομμύρια. Σύνολο 272. 130 είναι από τους έμεσους φόρους, ΦΠΑ και το φόρο κατανάλωσης 100. Για να έχετε μια ιδέα πώς έχουν οι φόροι μας, κυρίως από εμέσους φόρους έχουμε εισόδημα. Από το 2013 αποφασίσαμε να ε, διευκολύνουμε την κατάσταση γιατί είχαμε συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης. Και για τα, κατά τα άλλα είναι ένα πιο μικρό τμήμα, αλλά αυτό είναι από τις εταιρείε κυρίως στις τράπεζες. Και από τους ξένους είναι οι φόροι το μη κατοίκων. Μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία για να έχετε κάποια ιδέα. Και προφανώς δεν το κάνουμε για τους φόρους που έχουμε αυτές τις συμφωνίες. Θέλουμε να διαφοροποιήσουμε την οικονομία μας, γι' αυτό το κάνουμε. Και να μην έχουμε μόνο τους παραδοσιακούς τομείς αλλά και νέους τομείς όπως της υγείας, πληροφορική και άλλα που συνδυάζονται και με τον τουρισμό και με τους επισκέπτες μας. Αυτό θέλουμε, να διαφοροποιήσουμε την οικονομία μας και να την μεγεθύνουμε. Δεν ξέρω αν σας βοηθάνε αυτά από παντού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Συμπληρωματική ερώτηση προς τον εκπρόσωπο του Μονακό, θέλω να ρωτήσω πώς εφαρμόζεται αυτό τον καιρό την πρωτοβουλία BEPS του ΟΣΑ πρώτον. Δεύτερον, τι κάνετε για τις εκθέσεις αναχώρα ε, για ε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τρίτον, τι λέτε για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και για τις φορολογικές συμφωνίες, ε, tax rulings και ε, προκαταρκτικές ε, συμφωνίες. Ευχαριστώ, υπουργό. Έχω και πάλι την εντύπωση ότι τοποθετήθηκα για αυτό το ζήτημα, αλλά με τα χαρά να απαντήσω και πάλι και θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο για τις φορολογικές ε, συμφωνίες. Για τον ΠΕΠΣ, στις ε, επόμενες εβδομάδες και μήνες θα εξετάσουμε τις νέες εξελίξεις. Ε, σας εξήγησα για ποιο λόγο δεν το έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Και στο, στις 22 Φεβρουαρίου στο Μονακό το συζητήσαμε και με τον κύριο Μοσκόβηση. Όπως είπανε, και άλλοι για την έκθεση, υποβολή εκθέσεων αναχώρα θα πρέπει να το συζητήσουμε λεπτομερώς και όποια μέτρα κρίνουμε απαραίτητα θα τα αναλάβουμε αμελητή όπως και οι υπόλοιποι συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία δεν μιλάμε για κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε για τρίτες συνδεδεμένες χώρες όπως και το πριγκιπάτο του Μονακό. Για τις φορολογικές συμφωνίες, ε, ο διευθυντής μας ε, για τις φορολογικές υποθέσεις θα ξαναπάρει το λόγο. Ε, για να μην υπάρξει παρανόηση, τι είναι η φορολογική συμφωνία. Ε, πρόκειται, υπάρχουν δύο είδη. Υπάρχουν οι αποφάσεις ερμηνείας Δηλαδή, όταν ε, μέσα σε 30 ημέρες λαμβάνει απάντηση στα ερωτήματά του κάθε φορολογούμενος. Δε, rulings δεν έχουμε, δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται. Mm. Έχουμε ένα παραδοσιακό φορολογικό σύστημα που ε, προσωμιά στο γαλλικό ε, δεν έχουμε ruling, δεν, δεν υφίσταται, δεν προβλέπεται στην νομοθεσία μας. Mm. Ε, ε, άρα, στην ΤΑΞ 1, την Προσωρινή Επιτροπή, πέντε μήνες εξετάσαμε το θέμα και είδαμε, για να τα πούμε απλά, ότι υπάρχουν δύο είδη ε, ρεσκρί στα γαλλικά και ruling στα αγγλικά. Αλλά το ruling είναι η μετάφραση του ρεσκρί. παρότι συμπίπτουν οι όροι, είναι δύο διαφορετικές πρακτικές. Ε, η φόρμουλα, είτε ρεσκρή είτε ruling υπάρχει σε όλες τις χώρες και ποιο είναι το ε, μεγάλο πλεονέκτημα για το φορολογούμενο. Είτε είναι ιδιώτης, είτε ηθικό πρόσωπο, ίδρυμα, ε, ένωση, σωματείο, ε, ε σωματείο, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο είναι. υπάρχει μια σιγουριά για το φορολογικό καθεστώς που θα εφαρμοστεί στη δική του περίπτωση. Εκεί όπου έχει την έδρα του. Όταν ανοίγει κάποιο τα βιβλία του ή αλλάζει καθεστώς ε, ή είναι ε, έχει την έδρα του ήδη σε, αυτό το, σε αυτή τη χώρα, σε αυτό τον τόπο, αλλά έχει ε, ερωτήσεις για την έμεση, την άμεση φορολόγηση, για την καταχώρηση των Μητρώων, παραδείγματος χάρη, έχει τη δυνατότητα να αποταθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή και να υποβάλει το ερώτημα σε σχέση με το εφαρμοστέο φορολογικό καθεστώς. Ε, κατά τη γνώμη μου εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται παραδείγματος χάρη ο ΦΠΑ ή δεν εφαρμόζεται ο εταιρικός ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων ποιο είναι το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην περίπτωσή μου υποχρεούται γραπτός να απαντήσει η αρμόδια φορολογική αρχή και αυτή η απόφαση, αυτή η απάντηση έχει πολύ σοβαρές νομικές επιπτώσεις εάν ε, κάνει λάθος κατά την ερμηνεία του νόμου εις βάρος του κράτους η φορολογική αρχή υπερισχύει της κείμενης νομοθεσίας η απάντηση, γραπτή απάντηση αυτή. Είναι κατοχήρωση ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του φορολογουμένου. Όχι σε όλες τις χώρες. Στη δική μου 15 με 17.000 τέτοιες ε, φορολογικές αποφάσεις εκδίδονται ετησίως ε, και εφαρμόζονται με ικανοποιητικό τρόπο. Για διάφορα φορολογικά καθεστώτα σε άλλες χώρες διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ε, μεγαλύτερο περιθώριο ερμηνείας και κάποια ρεσκρή ή rulings ε, συνοδεύονταν από γραπτές συμφωνίες που περισσότερο ή λιγότερο πηχούνταν σε αυτές τις ε, γραπτές ε, συμφωνίες και απαιτήθηκε να τροποποιηθούν αυτές οι απαντήσεις για να υπάρξει μόρφωση τόσο ε, προς τη στάση του ΩΣΑ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θετήσαμε στο τέλος του 2014 μια σχετική έκθεση και πέρα από τις συστάσεις ε, υπάρχει πίεση από την κοινή γνώμη για την ε, ολική διαφάνεια και φορολογική δικαιοσύνη. Αυτή η πίεση απορρέει από ε, αριθμό σκανδάλων που έκαναν τον πάταγο που ξέρουμε όλοι, όπως το LuxLeaks. Θα σας πρότεινα να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά αυτό το γύρο των ερωταπαντήσεων. Ε, ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους ε, των τριών χωρών που ήρθαν στη σημερινή ακρόαση. Νομίζω η συζήτησή μας ε, περιστράφηκε γύρω από τα θέματα διαφάνειας και του εταιρικού φόρου. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, θέλω μόνο να πω ότι όντως διαπίστωσα ότι έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση Έχουμε ε, στις συμφωνίες ε, τις φορολογικές την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ε, ανάμεσα στην Ένωση και τις χώρες σας. Όμως ε, έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε με το Liechtenstein. μιλήσαμε για τα ιδρύματα και τα καταπιστεύματα. Γι' αυτό το ζήτημα είναι ξεκάθαρο ότι χρησιμοποιούνται για φορολογικό σχεδιασμό από τις πολυεθνικές ε, αυτά τα ιδρύματα στο Λίχτενστάιν. Είναι παγκοσμίως γνωστό, ε, ε, ασχέτως με αυτά που μας είπατε. Ξέρουμε τι γίνεται με τα ιδρύματα, με την, το δικτωσιακό καθεστώτος των επιχειρήσεων και τα τράσεις. Για την εφαρμογή τώρα των πρωτοβουλειών ΟΣΑ και BEPS, Πρέπει να, δούμε, να διαπιστώσουμε, επιθυμείτε ε, τη διαφάνεια. Αν ναι, θα πρέπει να περάσετε σε ένα σύστημα πολύ εκθέσεων αναχώρα. Είναι ένα από τα πολύ σημαντικά εργαλεία που εξασφαλίζουν ε, την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Για την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση, σε συζητητή, η BIM, θα προκύψει αυτό το θέμα με ιδιαίτερη ένταση αργότερα το 2016, χρειαζόμαστε κοινή προσέγγιση. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, να σε ευχαριστήσω θέλω που ήρθατε και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τους προσκεκλημένους μας για όλες τις απαντήσεις που έδωσαν τους εισηγητές, τα μέλη της Επιτροπής και να αναφέρω πώς Το καταλάβατε εξάλλου γιατί υπενθυμίσατε και ότι έχουν καταβληθεί πολύ σημαντικές προσπάθειες ε, του, τα περασμένα χρόνια. Λοιπόν, θα έχετε καταλάβει ότι για τον εταιρικό φόρο, γιατί είναι η ε, ε, μοναδική μας αρμοδιότητα εδώ σε αυτή την προσωρινή επιτροπή, να σημάνουμε μια νέα εποχή. Η εποχή όπου γινόταν αποδεκτή αυτή αποδεκτός αυτός ο φορολογικός ανταγωνισμός ε, των κρατών με άνισους όρους ανταγωνισμού, αυτή η εποχή έχει παρέλθει. Ε, όπως επίσης η εποχή του ε, τραπεζικού απορρίτου έχει ε, εξίσου παρέλθει. Και γνωρίζετε όλοι πως κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες που για ιστορικούς λόγους βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη κατάσταση πολιτικής με αναξαρτησίας αλλά ιδιαίτερη ισχυρής οικονομικής εξάρτησης από τις γειτονικέ χώρες ε, ε, εποφελήθηκαν από αυτό το φορολογικό ανταγωνισμό, τον αθέμητο φορολογικό ανταγωνισμό. Παρήλθε αυτή η εποχή όπως σας είπα. Επανάσταση δεν θα γίνει εν μία νυχτή, όμως θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις και θα πρέπει να ξέρετε πως το Κοινοβούλιο παρέτεινε την εντολή της ε, προσωρινής επιτροπής για το ίμιση, μέχρι το ίμιση του 2017 και όπως σήμερα θα προβούμε στην εξακρίβωση μόρφωσης με αυτές τις συστάσεις που κάνουμε, τις ε, διεθνείς συμφωνίες, συμβάσεις που έχουν υπογραφεί και ιδιαιτέρως ε, για τις ε, προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν τον Ιανουάριο του 2016 για την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΣΑ κατόπιν. θα υποβάλει συστάσεις ε, η Επιτροπή μας ε, για την, ε, το περίφημο CCCTB, είναι το ακρονίμιο για την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση. Θα υποβάλουμε λοιπόν συστάσεις και για αυτό το θέμα. Κατόπιν έχουμε το σχέδιο BEPS στο ΩΣΑ και θα ακολουθήσουν και άλλες συστάσεις από εμά ε, ε, και οι φορολογικές αρχές ε, ανά τον κόσμο, αυτός είναι ο στόχος, θα εφαρμόσουν τις συστάσεις. Φυσικά ουτοπιστές δεν είμαστε. Θα είναι δύσκολη, επαχθή διαδικασία και χρονοβόρα. Παρ' όλα αυτά, ξεκινούμε και αναλαμβάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση τρεις πρωτοβουλίες ε, για να ενισχύσουμε την εφαρμογή και για να ε, κάνουμε ε, τις δράσεις που απαιτούνται. Έχουμε από τα 28 κράτη-μέλη προσώπους κοινοβουλίων ε, που θα έρθουν στις 17 Απριλίου για τις ε, ε, προτάσεις, συγγνώμη, στις 18 Απριλίου για τις προτάσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το ζήτημα. Αυτό το κάνουμε με στόχο να εκπονήσουμε και εμείς τις συστάσεις μας που εγκρίναμε και που ε, χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 18 ε, ε, Απριλίου, λέει ο πρόεδρος, τώρα είναι η εκπρόσωποι των Υπουργών Οικονομικών και όχι των Κοινοβουλίων. μετά, στην έδρα του ΩΣΑ συνάντηση με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων όλων των χωρών που στα πλαίσια του ΟΣΑ συμμετείχαν στην εκπόνηση σχεδίου δράσης. Και εσείς φυσικά συμμετείχατε και κατά πάσα πιθανότητα θα σας προκαλέσει όσα. Πάνω από 80 χώρες δηλαδή συμμετείχαν. Ίσως δεν έχουμε τους εκπροσώπους των κοινοβουλίων ε, των 80 χωρών, αλλά θα εκπροσωπηθούν όλων των ειδών οι χώρες, όχι μόνο οι πλούσιες, όχι μόνο οι G20, ε, θα έχουμε εκπροσώπους από όλες τις χώρες, από όλες τις υπήρους, αν ε, προηγουμένου, για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Είναι ε, ορόσημο για την μετάβαση σε ένα διαφανέστερο και δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Το δεύτερο ήμιση του Μαΐου θα πάει ε, μεταβεί στη, σε, είπα, μια προσωπία της Επιτροπής μας ε, για να ε, συνεργαστούμε με το Κογκρέσο της ΕΠΑ, τις δύο συναρμόδιες ε, επιτροπές. Λοιπόν, και θα συνεχιστούν οι εργασίες που προτείναμε, η συνεργασία μαζί τους, πρόσφατα γεγονότα όπως απόφαση μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων να μεταφέρουν την, έδρα τους, όχι μόνο να δημιουργήσουν μια θηγατρική, αλλά μεταφέρουν την έδρα τους από τις ΣΥΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε μεγάλη εντύπωση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ περνούν προεκλογική εκστρατεία και το θέμα τους ενδιαφέρει πάρα πολύ υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Και είναι σημαντικότατο για μας στα πλαίσια του ΟΣΑ, η της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να μην είναι οι μόνες μαζί με εσάς να εφαρμόσουν τις ε, συστάσεις του ΩΣΑ. Οι μεγάλοι εταίροι μας στον κόσμο θα πρέπει να κάνουν το ίδιο, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ. Και πρέπει να ασκήσουμε πειθό, διότι πρώτη ευθόρμητη αντίδραση του Κογκρέσου θεωρεί ότι δεν, ε, δεν υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση, δεν στηρίζει ιδιαίτερα τον ΩΣΑ και δεν αντιδρά θετικά το Κογκρέσο όταν τρίτες χώρες θέλουν να τοποθετηθούν όσον αφορά το δικό τους φορολογικό σύστημα. Κάθε μία από τις χώρες μας, καθένα τα πριγκιπάντα σα, τι χώρες είτε είναι δημοκρατία ή είναι πριγκιπάτο, είναι βασίλειο, θέλει να έχει την κυριαρχία όσον αφορά τη φορολογία. Λοιπόν, πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το θέμα και από την άλλη πλευρά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση Έχουμε και κάποιους οικονομικούς φορείς που έχουν παγκόσμιο μέγεθος και τζίρο που ξεπερνά το ΑΕΠ των περισσότερων χωρών του κόσμου και έναντι αυτό δεν μπορούμε να δρούμε με κατακαιρματισμένο τρόπο με αποτελέσματα δέχεται κοινή γνώμη. Σε αυτό το πνεύμα εργαζόμεθα και σε αυτό το πνεύμα προτείνω να συνεχιστεί η συνεργασία μας και σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά που ήρθατε εδώ σήμερα το πρωί. Λοιπόν, πέρας διακόπτεται η συνεδρίαση. Στις 3 η ώρα θα τα ξαναπούμε. Γεια σας και καλή όρεξη.